Uh, so good afternoon, everybody. Um, welcome to our meeting this afternoon. Καλό απόγευμα. Καλώς ήρθατε στην απογευματινή μας συνεδρίαση. Καλώς ορίζω και αυτούς που μας ακούν από το διαδίκτυο. Να σας ε, θυμίζω ότι όσοι ακούν από το διαδίκτυο θα έχουν ε, σύντομα και ένα newsletter το οποίο θα είναι προσβάσιμο από τον ιστότοπο της ε, Επιτροπής μας και για πρώτη φορά θα ε, περιλαμβάνει και αναφορά για τις διαδικασίες πρώτης ανάγνωσης. Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε τέσσερα σημεία στην ημερήσια διάταξη σήμερα το απόγευμα. Αφορούν γνωμοδοτήσεις, αλλά είναι παρόλα αυτά πάρα πολύ σημαντικά. Πρώτο θέμα είναι η πρόσβαση των προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων χωρών στην εσωτερική αγορά τη Ένωση στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. Πρόκειται για ένα σημαντικό θέμα, το οποίο εντάσσεται στη γενικότερη συζήτηση για τις δημόσιες συμβάσεις. Παρεμβάσει εκτό μικροφώνου, οι διερμηνεί δεν ακούν δυστυχώ. Ναι, το ονόμα σα συμμετρικό. Η είναι ο κύριος Φρανκ Έγγελ και είναι και σκιώδης ε, εισηγητής ε, για την ε, οδηγία για το δημόσιες συμβάσεις. Δεν είναι εδώ δυστυχώς σήμερα, αλλά έχουμε την κυρία Μπάρμπαρα Βάιλερ, η οποία είναι εισηγήτρια, συγγνώμη, σκιώδης για το τους σοσιαλιστές και είμαι και εγώ εδώ θα δώσω αμέσως το λόγο στον ε, συνάδελφο Σφάμπ για να ξεκινήσει την συζήτηση, να μας πει πώς ε, προτίθεται ο κύριος Έγγελ να προχωρήσει με την εργασία αυτή. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η γνωμοδότηση της Επιτροπής μας για την αρμόδια επί της ουσίας Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου έχει σαν αντικείμενο το πώς μπορεί μακροπρόθεσμα να διαμορφωθεί η εμπορική τοποθέτηση της Ευρώπης έναν των τρίτων κρατών. Υπάρχουν λοιπόν δύο διαφορετικές σχολές εδώ. Άλλοι λένε ότι πρέπει να παραμείνουν ανοιχτέ οι αγορέ ανά τον κόσμο, γιατί εμεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με τι ε, μεσαίε επιχειρήσει μα που στρέφονται προ εξαγωγέ έχουμε μέγιστο συμφέρον να παραμείνουν ανοιχτέ οι διεθνεί αγορέ και προσβάσιμε. Ενώ κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι θα πρέπει στην Ευρώπη να εισαχθούν μηχανισμοί οι οποίοι θα μπορούν να αντιμετωπίσουν άλλες δυνάμεις εμπορικές, οι οποίες δεν είναι τόσο πολύ ανοιχτές στις τάσεις του εμπόριο, ή να τις υποχρεώσουν να αποδιαρθρώσουν εμπορικούς και μη φραγμούς στο εμπόριο. Ε, δεσμολογικούς και άλλους φραγμούς στο, εμπόριο. Έτσι λοιπόν, στόχος εδώ του εισηγητού είναι να ε, βρει μια συμβιβαστική πρόταση. Ο κύριος Έγγελ δυστυχώς δεν μπόρεσε να είναι σήμερα εδώ. Εγώ προσπαθώ να εκθέσω τις θέσεις του. Επί της ουσίας δεν συμφωνούμε σε όλα τα θέματα, πρέπει να πω. Υπάρχουν και στο δικό μας, στη δική μας την ομάδα κάποιες ε, προτάσεις που να συζητηθούν. Η... Επιτροπή μας έχει μόνο ε, αγνομοδότηση, δυνάμει του άρθρο 50, αλλά θέλουμε να προτείνουμε την ε, ε, αναφορά στα ε, έντυπα και τους όρους του άρθρου 17.3 του, της διαδικασίας για, την, για τις αρμοδιότητες και το άρθρο 20 του, της προτάσεως του κανονισμού για τα άρθρα 85 και 90. Και υπάρχει μια σειρά από άρθρα, όπου έχουμε μαζί με την ίντα κοινέ αρμοδιότητε, το άρθρο 2, το άρθρο 7, άρθρο 2 για τους ε, ορισμούς, άρθρο 7 για τις ε, κατώτατε προτάσει. προσφορές, τη διαδικασία της Επιτροπής, το απόρριτο, την εισήγηση, το άρθρο 19. Και όπως είπαμε, Έχουμε συστήσει με τον κύριο Έγγελ την ε, τοποθέτησή μας ότι θα έπρεπε η Επιτροπή μας να έχει περισσότερες αρμοδιότητες. Ένα θέμα που επεξεργάζονται από κοινού η Επίτροπη Μπαρνιέ και Ντεγκιούχτ τελικά έχει πάρει, έχει προσλάβει διαστάσεις περισσότερο διεθνούς εμπορίου. Εξού και υποχρεούμαστε και εμείς να ακολουθήσουμε αυτή τη διαδικασία. Περαιτέρω συζητήσεις οι αναμενόμενε περαιτέρω συζητήσει με την αρμόδια του ΣΥΑΝ. Επιτροπή δεν φαίνεται να μας ε, δίνουν πολλά περιθώρια για ελπίδες. Εν πάση περιπτώσει θα μπορούσαμε για τον προσδορισμό της ε, προελεύσεω να έχουμε συζητήσει περισσότερο. Μπορούσαμε να κάνουμε επί παραδείγματι την παραπομπή στον τελωνιακό κώδικα. Και αυτό όσον αφορά τις αρμοδιότητες και τώρα θα περάσω στην κύρια πρόταση, στην ίδια την χρηματοδότηση. Έχουμε 0,08% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο διεθνές εμπόριο για λόγους ότι η πρόσβαση στους, στις διεθνείς ε, ε, αγορές είναι περιορισμένος ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει για τους ξένους ανταγωνιστές, για τα, τρίτα κράτη, ανοιχτή την ε, αγορά της, οι τρίτες χώρες δεν ακολουθούν την ίδια στάση. Και έτσι στις δημόσιες αγορές έχουμε πρόβλημα πρόσβασης. Άρα μπορούμε να διαπιστώσουμε δυναμικό μεγάλο, εφόσον ανοίξουν βέβαια οι αγορές των δημοσίων ε, συμβάσεων ε, των τρίτων κρατών. Έτσι λοιπόν. Για να αντιμετωπιστεί αυτή η ανισότητα, ανοιχτές αγορές Ευρωπαϊκής Ένωσης για, τρίτες, ε, για ενδιαφερομένους ε, τρίτων χωρών στις δημόσιε συμβάσει και αντίστροφα κλειστές αγορές των τρίτων κρατών, πρέπει να αξιοποιηθούν τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας ε, το μέσον το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει δεν πρέπει να μετατραπεί σε έναν τίγρη χωρίς δόντια, όπως λέει ο κύριος Έγγελ. Πρέπει δηλαδή να φέρει αποτελεσματικές λύσεις χωρίς ε, παρατράγουδα, χωρίς δηλαδή παρεπόμενες συνέπειες που θα μπορούσαν να αποβούν εις βάρος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα σήμαινε ουσιαστικά τι είδους δυσκολίες μπορούμε να περιμένουμε και για ποια περιοχή της Ευρώπης ε, εάν κάναμε την παρέμβαση αυτή με, το, με την πρόταση αυτή για το νομοθέτημα. Και περιμένω να ακούσω τις προτάσεις των συναδέλφων και τις ιδέες τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe... Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι πρέπει να μιλήσουμε όχι μόνο για τα αγαθά που θα εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τα ευρωπαϊκά αγαθά τα οποία θα πρέπει να εξάγονται σε άλλες χώρες. Και όπως είπε και ο κύριος Σβάμπ, η αγορά μας είναι σχετικά ανοιχτή, οι αγορές μας είναι σχετικά ανοιχτέ. Εάν θέλουμε λοιπόν εξελίξεις για τα επόμενα χρόνια και ανεξαρτήτως του πώς θα διαμορφωθεί η δημοσιονομική κρίση πάλι δεν πρόκειται να ξανακλείσουμε τις αγορές μας γιατί μου φαίνεται παράλογο μου φαίνεται αντίκθετο με, τις, με τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μου φαίνεται πολιτικά παράλογο να προσπαθούμε να διατηρήσουμε μια κατάσταση η οποία έχει Μα έχει οδηγήσει αυτό το σημείο, δηλαδή να, να συνεχίσουμε χωρίς καμία αλλαγή, να βρισκόμαστε στην ε, κατάσταση που εμεί έχουμε αγορέ ανοιχτέ, ενώ οι άλλοι όχι. Λοιπόν, πρέπει να δούμε... Ε, πρέπει να δούμε τα προϊόντα μας πώς μπορούν να φτάνουν και σε αναπτυσσόμενα κράτη. Πρόκειται δηλαδή, γιατί δεν μιλάμε μόνο για αναπτυσσόμενα κράτη, έχουμε να κάνουμε και με κράτη μεγάλο όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς που βρίσκονται σε ισότιμο επίπεδο. Δεν προσπαθούμε δηλαδή να πουλήσουμε προϊόντα στα πιο φτωχά κράτη της Αφρικής ε, ή όπου αλλού στον κόσμο. Αυτό είναι το πρώτο σημαντικό. Το δεύτερο είναι ότι ίσως θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας εξηγήσει ακόμη περισσότερο, γιατί δεν κατάλαβα ακόμα Εάν υπάρχει κάποια αντίφαση, ως προς τη ρύθμιση για τις ε, συμφωνίες GPA και αν υπάρχει ένα περιθώριο να τις βελτιώσουμε αυτές τις ε, συμφωνίες. Ή εάν υπάρχει περιθώριο να βελτιώσουμε κάτι σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, πρέπει να ρωτήσουμε εάν αρχίσουμε να διαπραγματευόμαστε σύμβαση ε, η εταιρική σχέση ελεύθερων συναλλαγών με τις ΗΠΑ, τι νόημα έχει να συζητούμε αυτή την προκείμενη πρόταση νομοθεσίας. Δεν καλυπτόμαστε από μια συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών ή αντίστροφα τι χρειαζόμαστε την FTA, τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών, εάν πρόκειται να εισαχθεί αυτό το ε, νομοθέτημα. Επίσης ε, θα ήθελα να ρωτήσω πού βρίσκονται τα όρια, πού βρίσκονται τα όρια σε σχέση με τα, με τρίτα κράτη. Και στο προτελευταίο μου σημείο τα θέματα τα οποία έχουμε να συζητήσουμε και να διαπραγματευτούμε με την Επιτροπή Εξωτερικού Εμπορίου, κύριε Σφάπ. Είναι αυτά βεβαίω που αναφέρατε πλην όμω εγώ θα ήθελα να υπογραμμίσω ένα πράγμα και πρέπει να πω ότι αισθάνομαι υπερήφανη που εμεί εδώ έχουμε μπορέσει να περάσουμε τι θέσει μα για τι άλλε νομοθεσίε σχετικέ με τι δημόσιε προμήθειε. Ε, το άρθρο 7 με τι abnormally low tenders, με τις ε, αφύσικα ε, χαμηλές προσφορές, κάτι το οποίο έχουμε να κάνουμε, έχουμε αντιμετωπίσει με Ρώσους και άλλα κράτη, δηλαδή ε, προτάσεις οι οποίες φαίνεται να είναι τόσο χαμηλές ώστε βρωμάνε κρατική επιδότηση. Και μάλιστα από κράτη που δεν είναι μόνο πολύ φτωχά, όχι μόνο από κράτη που είναι πολύ φτωχά σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και από κράτη πλούσια όπως η Ιαπωνία και άλλα. Άρα οι άκρως αυτές ε, χαμηλής αξίας προσφορές είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να προβλέψουμε, πρέπει να επιμείνουμε, πρέπει να υποστηρίξουμε και διαδικαστικά είναι όντως ε, σαφές ότι δεν έχουμε πολλές αρμοδιότητες και μάλιστα δεν έχουμε και κοινέ αρμοδιότητες, αλλά είναι τόσο σημαντικό αυτό το θέμα, γιατί είναι αχαρτογράφητο πεδίο, ε, το συγκεκριμένο. Ένα θέμα που άλλωστε θα έπρεπε να ανήκει στην Επιτροπή Βιομηχανία και δεν, το ήθελε. Ένα θέμα λοιπόν το οποίο θα μας φέρει αντιμέτωπος με τόσα θέματα βασικά της πολιτικής μας και επιλογές πολιτικές που είναι πιστεύω πολύ καλό το να εμπλακεί η Επιτροπή μας, όχι τυπικά έστω δεν είναι δυνατόν αυτό, αλλά πάντως άτυπα και ε, αφόρμητα ανεξαρτήτως του τι θα πει η Επιτροπή Εμπορίου εξωτερικό εμπόριο. Είχα παρακολουθήσει μια ακρόαση, αλλά ασφαλώ θα γίνουν και άλλες. Είναι πολύ περίπλοκο το θέμα και θα χρειαστεί να προσκαλέσουν και άλλους εμπειρογνώμονε. Ε, έτσι λοιπόν νομίζω ότι έστω και άτυπα πρέπει να είναι παρόντες οι εκπρόσωποι μα, οι σκιώδεις μα για το θέμα αυτό, ώστε να το παρακολουθήσουμε από κοντά. ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα, να πω ότι και εγώ συμφωνώ με τον κύριο Σφάμπ ότι βλέπουμε δύο τελείω διαφορετικέ σχολέ εδώ. Δεν ε, νομίζω ότι κανείς ε, μπορεί να αμφιβάλλει για το ποια σχολή εκπροσωπώ εγώ επί του θέματος αυτού. Πρώτον, να καταστήσω σαφές ότι συμφωνώ απολύτως ότι θα πρέπει να έχουμε σε εταίρους στι τρίτης χώρε και βεβαίω θέλουμε να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις όπου είναι εύκολη η πρόσβαση των ε, εταιριών μας, των επιχειρήσεών μας στις τρίτες χώρες. Πιστεύω, πιστεύω ακόμα ακράδαντα στην ελεύθερη αγορά. Και βεβαίως ε, θεωρώ ότι ε, θα πρέπει να δώσουμε μεγάλη σημασία και να υπογραμμίσουμε την αμοιβαιότητα Ε, να μην, ε, όχι να μην ανοίξουν ε, στον ανταγωνισμό οι ανοιχτές, οι κλειστές αγορές. Αντίθετα, δεν είναι δυνατόν να κλείσουμε τις αγορές μας, γιατί ούτως ή άλλως αυτό θα οδηγήσει σε διοικητικό άκθος, αλλά και αύξηση του κόστους. Για την πρόταση έχουμε μία συγκεκριμένη βάση. Ακόμα και η ίδια η Επιτροπή ε, για που ήταν υπεύθυνη για την ε, μελέτη αντικτύπου της ίδιας Επιτροπής ε, απεφάνθη ότι παραμένει πάρα πολύ ασθενής η θέση των εταιριών και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το ρωτήσουμε και στην Κομισιόν. Ε, έρχεται από την ίδια την Επιτροπή αυτή η διαπίστωση, να μας πει πώς προέκυψε η διαπίστωση αυτή. Επίσης ε, και η ε, Ακαδημία έχει εκφραστεί αρνητικά σε σχέση με την ε, πρόταση της ε, ε, Κομισιόν και εν πάση περιπτώσει με αυτά δεν μπορούμε να επιτύχουμε την ισορροπία την οποία ευαγγελιζόμαστε. Εγώ χρειάζομαι συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία για να πιστώ. Ίσως θα πρέπει λοιπόν πρώτα απ' όλα να μιλήσουμε με τους ανθρώπους οι οποίοι έκαναν αυτή την έρευνα και κατέληξαν σε αυτά τα αποτελέσματα. Επομένως είναι αμφισβητήσιμη όλη η βάση, η ίδια μάλλον η βάση ε, στην οποία έχει βασιστεί αυτή η πρόταση. Απ' την άλλη θέλουμε ενιαία αγορά. Να σας πω, ε, στο Λονδίνο μπορεί ε, να ε, απορριφθεί στο Λονδίνο, ενώ αντίστοιχα κινέζικα, κινέζικες προτάσεις μπορεί να γίνουν δεκτές στην Ισπανία ή στην Γαλλία. Στο άρθρο 6 νομίζω παραμένει και ένα μεγάλο πρόβλημα γιατί λέμε ότι υπάρχει δυνατότητα αποκλεισμού των προσφορών ε, επιδημοσίων συμβάσεων ε, βάσει κρίσης των τοπικών παραγόντων. Η πρότασή μου νομίζω είναι να διαγραφεί το άρθρο 6 και να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στα άρθρα 8 μέχρι 11 και η Κομισιόν να ξεκινήσει διαβουλεύσεις και συζητήσεις με ε, τα ε, κράτη αυτά τα οποία περιορίζουν την πρόσβαση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. η Κομισιόν ας πούμε έχει ε, ξεκινήσει συζήτηση με την Βραζιλία όσον αφορά την άρση προσκομμάτων για την συμμετοχή σε δημόσιες συμβάσεις και την ίδια ώρα η Δανία αποκλείει ε, προσπάθειες της Βραζιλίας να πάρει δημόσιες ε, συμβάσεις. Ναι. Είμαι σίγουρος ότι συμφωνούμε όλοι ότι θέλουμε περισσότερες αγορές δημοσίων συμβάσεων και αυτό έχει να κάνει με το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας και νομίζω ότι αυτό τουλάχιστον είναι ένα σημείο επί του οποίου συμφωνούμε όλοι. Αυτά για την ώρα. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ρούλα. Θα ξαφνιάσω τον πλωρολίστατα, αλλά συμφωνώ με όλα τα σημεία της αναλυσής του πλην ενός ότι εγώ καταλήγω στην ε, απόλυτη απόρριψη του κανονισμού γιατί είναι λάθος εργαλείο. Δεν μπορούμε να κάνουμε εμπορική πολιτική με τέτοια μέσα στις δημόσιες προμήθειες. Νομίζω ότι πρέπει να βρούμε λύσεις και σωστά λέτε ότι υπάρχουν αναλύσεις και από την Ευρωπαϊκή Επίτροπη επίσης βλέπουμε ότι οι δημόσιες προμήθειες μόνο 1,6%. Υπάρχει μαζί με τις θηγατρικές 15%. Δηλαδή στο χαρτί μπορεί να είμαστε μπορεί να έχουμε αγορέ αλλά στην πραγματικότητα είναι περιορισμένη η αγορά. Δεν είναι πρόσφαρη για μια εμπορική πολιτική πραγματικά. Και στο άρθρο 6 μπορώ να συμφωνήσω ότι βρίσκονται πράγματι σε πολύ δύσκολη θέση και αμηχανία οι μικρές επιχειρήσεις όταν, βρίσκονται, όταν καλούνται να αποφασίσουν για την ε, πολιτική αυτή για μια πολιτική που έχει συνέπειες και γραφειοκρατικές και σε κόστος και έτσι αντί να διευκολύνουμε την πρόσβασή μας στις αγορές τρίτων κρατών, μάλλον θα οδηγηθούμε στο αντίθετο αποτέλεσμα, στο μη επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, γιατί θα κλείσουμε κάποιους τομείς τελείως. Γι' αυτό απορρίπτουμε την οδηγία, λέει τώρα η ομιλήτρια, και έτσι κανονισμό, το χειρότερο είναι ότι είναι και κανονισμός, τουλάχιστον να ήταν οδηγία. Απορρίπτουμε λοιπόν τον κανονισμό και βλέπουμε ως προβληματικό ιδιαίτερα το γεγονό ότι επανέρχεται και ότι δυστυχώς όταν φτάνει πια στο κοινοβούλιο μια, απόφαση, μια πρόταση για να ψηφιστεί δεν καταφέρνει σχεδόν ποτέ το κοινοβούλιο να την απορρίψει απλά και μόνο. Γι' αυτό βασικά απευθύνω έκκληση προς το Συμβούλιο. Νομίζω ότι η κυρία Μακλάρκιν δεν είναι εδώ. θέλετε εσείς να παρέμβετε εξ ονοματός της. Πολύ ωραία λοιπόν, γιατί διαφορετικά θα, τα, θα αναλάβανα εγώ το βαρύ αυτό έργο. Θα μιλήσω εξ ομένως της κυρίας Έμα Μακλάρκιν. Είναι σημαντική η συζήτηση αυτή στην Επιτροπό ε, ΙΜΠΕ όσον αφορά ε, την ε, πρόσβαση προϊόντων και υπηρεσιών των χωρών στην εσωτερική αγορά της Ένωσης. Έχει συμμετάσχει στην αδελφό μου σε πολλές σχετικές συζητήσεις και κατέστησα φέσα ότι η συζήτηση δεν είναι ειλικρινής όπως αναφέρθηκε ήδη, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την σημασία αυτού του θέματος. 19% ε, του ε, ΑΕΠ αφορούν αυτές, ε, αυτά τα προϊόντα και οι υπηρεσίες τη στιγμή που διανύει ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές η Ευρωπαϊκή Ένωση και επομένως όταν μιλάμε για συμβάσεις δημοσίου, δημοσίου για δημόσιες συμβάσεις θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά αυτήν την δεν είναι ανάλογη με το διακύβευμα δεν ανοίγουν αρκετά οι τρίτες χώρες ε, την, ε, τις αγορές ε, για τις επιχειρήσεις της Ευρώπης και τελικά δημιουργείται πρόβλημα και κόστος για τους φορολογούμενους. Όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι, το άρθρο 6 είναι ένα πολύ σημαντικό άρθρο το οποίο δυσκολεύει. θα πρέπει να τροποποιηθεί αυτή η οδηγία το άρθρο 6 επιτρέπει με μονομένες ε, αρχές ή οντότητες των κρατών μελών να ζητούν από την Επιτροπή να εξαιρέσουν προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν ε, υφίστανται τους ε, κανόνες της πρόσβασης των διεθνών αγορών, αλλά αυτό μπορεί να αναφέρεται στο 50% των δημοσίων συμβάσεων η πρόταση αυτή ε, μας βάζει στον κίνδυνο να διακινδυνεύσουμε ε, πολλές ε, διακοπές εις την αλυσίδα εφοδιασμού και οπωσδήποτε πρόκειται και για νομοθέτημα το οποίο μπορεί να αποβεί πολύ επικίνδυνο για τις επιχειρήσεις μας Επίσης υπάρχουν και μακροπρόθεσμα ε, στοιχεία, ε, επιπτώσεις που μπορεί να έχει η εφαρμογή της οδηγίας στην αγορά. Μπορεί να βγουν από την αγορά κάποιες ε, επιχειρήσεις οι οποίες θα μπορούσαν να κάνουν πολύ καλές προσφορές όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις και θα συνέβαλαν στην πραγματική ολοκλήρωση της ε, αγοράς ε, και ε, οπωσδήποτε για μία ακόμα φορά θα την πληρώσει ο φορολογούμενος από τον οποίο θα αποστερήσει αυτή η διαδικασία πολλά χρήματα. Γι' αυτό λοιπόν ρωτώ την Επιτροπή τι θα συμβεί εάν η Επιτροπή Εσωτερικού Εμπορίου, Εσωτερικής Αγοράς ε, και η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου ε, καταλήξουν στο ίδιο αποτέλεσμα τι θα γίνει εάν ε, το Κοινοβούλιο αποφασίσει να μιλήσει με μία φωνή. Επίσης η συνάδελφος ε, θέλει να καταλάβει πώς θα λυθεί το πρόβλημα. Και επίσης ε, λαμβάνοντας υπόψη ότι στη νέα πρόταση αμοιβαιότητα συμπεριλαμβάνονται στοιχεία και ε, από τις δημόσιες συμβάσεις αλλά και από άλλα συναφή θέματα η αγορά δημοσίων συμβάσεων είναι ε, ανοιχτή όπως θα ήθελε να μας κάνει να πιστέψουμε η Επιτροπή ή ε, οι εκπρόσωποι τρίτων χωρών που συμμετέχουν ε, σε συμβάσεις έχουν τις ίδιες Ε, πραγματικά τις κερδίζουν ή απλό, έναντι τρίτων χωρών ή απλώς τις κερδίζουν επειδή ε, έχουν κάποιες ε, ιδιαίτερες στενές σχέσεις με τρίτες χώρες π.χ. με την Κίνα. Νομίζω ότι πιστεύουμε ότι αυτού του είδους συμφωνίες μπορεί να αποβούν εξαιρετικά καταστροφικές στις διμερείς σχέσεις ε, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτών των τρίτων χωρών. Ε, η κυρία Μαρκάρκιν ε, θεωρεί ότι με αυτό το κείμενο τελικά θα οπισθοδρομήσουμε και ελπίζει ότι στους επόμενους μήνες η συζήτηση θα βελτιώσει το κείμενο. Ευχαριστώ. Θέλει κάποιος άλλος να πάρει το λόγο, κυρία Στάιλερ, που δεν μιλήσατε. Όχι. Ίσως θα μπορούσα να κάνω κι εγώ ένα-δυο σχόλια. Οπωσδήποτε εγώ απολύτως ε, συμφωνώ με τους τρεις τελευταίους ε, ομιλητές, αλλά θα κάνω και κάποια ερωτήματα σαν πρόεδρος αν μου επιτρέπετε. Νομίζω, λοιπόν, και ως πρόεδρος το λέω αυτό, ε, η Επιτροπή μας χρειάζεται απαντήσεις. Πρέπει να απαντηθούν τα ερωτήματά της. Κυρίως θα ήθελα να έχουμε απαντήσεις από την Κομισιόν πάνω στο γεγονός, το συγκεκριμένο. Δηλαδή, Έχουμε σχεδόν ξεκινήσει ήδη διμερείς ε, διαπραγματεύσεις ε, με την Ιαπωνία και την, τις Ηνωμένε Πολιτείες που είναι βεβαίως πολύ σημαντικές ε, αγορές ε, δημοσίων ε, συμβάσεων, στις οποίες δεν έχουμε και μεγάλη πρόσβαση. Και νομίζω ότι αν συνεχίσουμε στο δρόμο που χαράζει αυτή η πρόταση, τότε θα συμπέσει με το άνοιγμα των ε, συζητήσεων για τις εμπορικές συμφωνίες και αυτό δεν είναι μια έξυπνη και σωστή επιχειρηματική κίνηση νομίζω από τη δικιά μας πλευρά. Θα ήθελα λοιπόν η Γενική Διευθυντή Trade να μας εξηγήσει πώς ε, το βλέπουν. Θα γίνει φασαρία, θα ακουστούν πολλά περί προστατευτισμού εάν προχωρήσει αυτή η πρόταση. Δεν θέλω να χάσουμε την ώρα μας εδώ, αλλά να μείνει στα συγκεκριμένα γεγονότα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να, να μας απαντήσει με συγκεκριμένο τρόπο. Πώς θα προχωρήσει λοιπόν με αυτό το κείμενο για τις δημόσιες συμβάσεις και πώς ταυτόχρονα θα φερθεί με αυτόν τον τρόπο σαν αφορά την πρόσβαση των τρίτων χωρών. Και κάτι άλλο για την οδηγία ε, περί δημοσίων συμβάσεων. Συζήτησα το θέμα με τον κύριο Μπαρνιέ. Και βεβαίως ε, είναι από τα λίγα σημεία επί των οποίων διαφωνούμε εντελώς με τον Επίτροπο Μπαρνιέ. Αυτή την ώρα υπάρχουν μεμονωμένες χώρες μέλη οι οποίες εφαρμόζουν την δικιά τους ε, ε, πολιτική. Αλλά αν θέλουμε πραγματικά να έχουμε ενιαία αγορά θα πρέπει να διατηρήσουμε και να συμφωνήσουμε μάλλον οι υπερηγών προνοιών και να συμφωνήσουμε όλοι. Δύο παρατηρήσεις από αυτού. Πρώτον, νομίζω ότι έχοντας πλέον και τα στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται στην μελέτη αντικτύπου και σε άλλες παρεμφερείς μελέτες, ότι εδώ έχουμε πρόβλημα γιατί όπως είπαν και οι τρεις προλύσαντες συνάδελφοί μου που βλέπουν με δυσπιστία την ε, ουσία και την αξία αυτής της πρότασης ε, αυτό καταδεικνύει και την ίδια μελέτη αντικτύπου. Αλλά πέραν αυτού είμαι σίγουρος ότι η Κομισιόν έχει κάποια εργαλεία έτσι ώστε να υπάρξει συμμόρφωση εν τέλει με τους κανόνες όσον αφορά και στα πλαίσια μάλλον τις παρούσες οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις. και το κατόφλι βέβαια είναι παρόμοιο με αυτό που προτείνεται εδώ φαντάζομαι. Επομένως, χρήσιμο θα ήταν εάν η Κομισιόν μπορούσε να μας εξηγήσει ποιο ήταν το πρόβλημα που προσπάθησε να λύσει με αυτήν την επιπλέον πρόσβαση όσον αφορά την ασύμβατη εφαρμογή της οδηγίας περί δημοσίων συμβάσεων. Συγκεκριμένες απαντήσεις αν είναι δυνατόν. Ε, υπάρχουν και κάποιοι συνάδελφοι οι οποίοι ενδεχομένως ε, βλέπουν το, την πρόταση με λίγο πιο θετικό βλέμμα. Εγώ πάντως είμαι εξαιρετικά δύσπιστος. Ε, με μεγάλο σκεπτικισμό τη βλέπω την πρόταση αυτή. Ο κύριος Πύρινος είναι εδώ από την Γενική Διεύθυνση Μάρκτ. Έχουμε και εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου, η Γενική Διεύθυνση Trade. Ποιος θέλει να ξεκινήσει. Thank you very much, Chairman. This is uh, Anders Jessen from DG Trade, for those who have not met. Από τη Γενική Διεύθυνση Εμπορία, για όσους δεν έχουν συναντήσει πιο πριν. Θα ήθελα λοιπόν ξεκινώντας να αναφερθώ στις πτυχές του άρθρου 6, ιδιαίτερα. Και για τις ερωτήσεις κυρίας Βάιλερ, αν υπάρχουν μέσα νομοθετήματα ήδη σε σχέση με τις, ε, τη συμφωνία με τις ε, κρατικές προμήθειες, με τις δημόσιες προμήθειες. Ναι, υπάρχουν, δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε κανέναν πέραν αυτής, της συμφωνίας GPA, ε, όπως αυτή κατέληξε μετά τις διαπραγματεύσεις πέρσι. Και έτσι, δεν έχουμε πολλέ προσδοκίε. Χρειάστηκαν άλλωστε πολλά χρόνια για να ολοκληρωθεί ο τελευταίο αυτό γύρο που κατέληξε στο GPA. Επομένω, τι έχουμε εδώ. Γιατί αυτό βλέπω να απασχολεί ε, ιδιαίτερα. Με ποιο πρόβλημα είναι αυτό που προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε. Λοιπόν, έχουμε μια σειρά από προβλήματα και δύο σχολές, θα έλεγα, ή και τρεις ακόμη, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπάθησε να κατευθύνει τις... Ε, ε, συστήσεις προ την χρυσή τομή, προς τη μέση οδό. Και όταν είχαμε ξεκινήσει το 2010 κάποιοι ζητούσαν να λάβουμε μέτρα αρκετά ριζικά, να κλείσουμε δηλαδή οτιδήποτε δεν έχει ακόμη ανοίξει και μόνο επιλεκτικά να ανοίγουμε τις δυνατότητες για χώρες οι οποίες θα ήταν διατεθειμένες να προσφέρουν αμοιβαία πρόσβαση μία λύση αυτή, ενώ κάποιοι άλλοι μας έλεγαν όχι μην πειράξετε τίποτα, μια χαρά είμαστε έτσι, περιοριστείτε μόνο στις διαπραγματεύσεις. Εμείς λοιπόν προσπαθήσαμε να χαράξουμε τη μέση εδώ, μία πρόταση και αυτό εδώ είναι μοναδικό πρέπει να σας πω στον κόσμο ολόκληρο, μια μοναδική ε, λύση που είναι η εξορισμού ανοιχτή αγορά. De jure μάλιστα, όχι de facto, εκ νόμου και δεν υπάρχει πουθενά άλλου στον κόσμο αυτό. Έτσι κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω πώς θα ε, αντιδράσουν οι εταίροι μας. Ούτε οι Ηνωμένε Πολιτείε ούτε η Ιαπωνία έχουν πάντω διαμαρτυρηθεί για την πρόταση. Και βέβαια ξέρουν πολύ καλά ότι έτσι έχουμε περισσότερη μόχλευση. Ε, θα προτιμούσαν ασφαλώ να μην είναι ε, τόσο δυνατή η θέση μας στις διαπραγματεύσεις, αλλά όπως και να έχει, ε, εμείς έχουμε αυτή τη θέση, ότι δηλαδή εξορισμού είμαστε στη διάθεσή τους για διαπραγμάτευση. Και βλέπουμε και από την προετοιμασία τους για τις διάφορες ε, προτάσεις και διαπραγματεύσεις ότι δεν εκφράζονται ούτε από τους Αμερικανούς ούτε από τους Ιάπωνες ανησυχίες ότι μπορεί με αυτόν τον πίνακα να διαταραχθεί η πορεία των διαπραγματεύσεων. Η δική μου η απάντηση ήταν «Ναι, είμαι βέβαιος, διότι αποστέλαμε διάφορες προτάσεις στα κράτη-μέλη και είχα διαπιστώσει ότι θα ήταν μάλλον, μάλλον ευχαριστημένοι αν βλέπανε μια θετική ανοιχτή στάση και αυτή τη μόχλευση από πλευράς μας. Επομένως αυτό που λέμε εμείς είναι η αδίποτε διεθνής μας ε, δέσμευση από συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών FTA ή από ε, τη συμφωνία ε, για τις δημόσιες προμήθειες, GPA, παραμένει ισχύ δεν ε, αντιμετωπίζει πρόβλημα και έχουμε ένα κεντρικό σύστημα που είναι θέλουμε να διαπραγματευτούμε πρόσθετη πρόσβαση. Θέλουμε την πρόσβαση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θέλουμε να κλείσουμε τις ευκαιρίες για πρόσβαση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν τα κοιτάξετε λοιπόν αυτά, η, πρόσθετη αυτή ε, επιλογή προκύπτει εφόσον προσδεριστεί μόνο όταν ε, διαπιστώσουμε σοβαρή και επίμονη διάκριση εις βάρον των δικών μας επιχειρήσεων, όταν ε, δεν οδηγήσουν πουθενά οι διαπραγματεύσεις ή όπου η χώρα μας αρνείται ακόμη και το διάλογο, τότε μόνο επιβάλλουμε την επέμβαση, αυτά τα περιοριστικά μέτρα. Το άρθρο 6 ε, δεν εφαρμόζεται καν στο όριο των 5 εκατομμυρίων. Είναι μια μονομερής δέσμευση για να είναι ανοιχτή η αγορά. Η κυρία Βάιλερ νομίζω επίσης ερώτησε αν έχουμε χάσει κάποιο τρένο. Όχι, δεν έχουμε χάσει κανένα τρένο. Διότι το καλοκαίρι, εφόσον μα δοθεί σχετική εντολή, σκοπεύουμε να αναπτύξουμε τι διαπραγματεύσει μα με τι ΗΠΑ. Ο Επίτροπο ήταν στην Επιτροπή Διεθνού Εμπορίου χτε, όπου εξέθεσε τις εξελίξεις. Όπου βέβαια ενδέχεται ε, να θεωρηθεί από τον εταίρο ως ε, δεδομένη η ανοιχτή μα στάση και όταν ε, προσπαθήσουμε ή επιδιώξουμε μια διαπραγμάτευση να μην κάνει καμία προσπάθεια. Ε, από την άλλη, εμείς έχουμε συστήματα ανοιχτά στις επενδύσεις. Έρχονται πολλές από τις εταιρείε αυτές ε, για επενδύσεις με ε, θυγατρικές όμως και πολλές φορές δεν καταγράφονται καν στις στατιστικές. Γι' αυτό θα προτιμούσα και εγώ κάποιοι από τους εταίρους μας, τους εμπορικούς, να προσέφεραν τις ίδιες ευκαιρίες για ε, επενδύσεις ε, στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις όσες προσφέρουμε και εμείς στις δικές τους. Δεν πάει τόσο, δεν έχουμε χάσει κανένα τρένο. Ήρθε η ώρα να, ε, έχουμε, να εξασφαλίσουμε ένα επιπλέον εργαλείο ώστε να δείξουμε ότι δεν πρέπει να μας θεωρεί κανείς δεδομένους. Θέλουμε να είμαστε ανοιχτοί βεβαίως, ή είμαστε δεθμένοι να μείνουμε ανοιχτοί βεβαίως, αλλά θέλουμε τις ίδιες ευκαιρίες και για τις δικές μας επιχειρήσεις. Για τις αναπτυσσόμενες χώρες και το όριο. Οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, LDCs, και οι υπηρεσίες τους και τα αγαθά τους καλύπτονται πλήρως, δηλαδή έχουν πλήρη πρόσβαση. Ούτε καν μπορεί να εφαρμοστεί σε αυτές το σχετικό νομοθέτημα. Έχουν μονομερή από πλευράς μας ε, ανοιχτή πρόσβαση. Οι αναδυόμενες οικονομίες φυσικά έχουν διαφορετική μεταχείριση και περιμένουμε να δούμε αν η Κίνα, η Ινδία ή άλλοι εμπορικοί εταίροι έχουν και για τις δικές μας ε, εταιρείε τη διάθεση να δείξουν ανοιχτό πνεύμα. Πάντως, θέλουμε σε μια εποχή μάλιστα δημοσιονομικής λιτότητας να ε, μην χρειαστεί να πιέσουμε ακόμη περισσότερο τις ε, ευκαιρίες τις οικονομικές που μπορούν να προσφέρονται και γι' αυτό και στο άρθρο 6 σημειώνουμε ότι δεν υπάρχει κανένας περιορισμός εφόσον θεωρεί μια εταιρεία ότι καλύπτεται επαρκώς, δηλαδή ότι ικανοποιείται οικονομικά. Το τι γίνεται τώρα γιατί με τις ε, δημόσιες αρχές που είναι οι κύριοι πελάτες, οι μεγαλύτεροι πελάτες κάποιων επιχειρήσεων και βλέπουν ότι στην Ευρώπη δύσκολα πια μπορούν να αναλάβουν συμβάσεις από το δημόσιο τομέα, θα τις βοηθήσουμε να αναπτύξουν τις δραστηριότητες τους και έξω από την Ευρώπη για να σταθούν στα πόδια τους. Φυσικά και ναι, και αυτό είναι το μέσο που προσπαθούμε να αναπτύξουμε ώστε να τους προσφέρουμε καλές ευκαιρίες και στο εξωτερικό. Αυτά νομίζω. Πιστεύω να έχω απαντήσει και στα κύρια ερωτήματα. Για το άρθρο 6 ιδιαίτερος. ευχαριστώ. Νομίζω ότι ο συνάδελφος ήδη πάρα πολύ καλά, σα ανέπτυξε τα επιχειρηματά μα, αλλά θα πρέπει εγώ να σταθώ σε κάποιε πηγέ του θέματο διότι όντω, αν κάνει ρίξει μια ματιά με ποιο τρόπο ε, έχει, έχει ε, δημιουργηθεί αυτό ο κανονισμός, ε, είναι κάτι το οποίο ακριβώ συνδέεται με τη φυσική και όχι μόνο αυτό, αλλά πρόκειται για ένα άνοιγμα το οποίο αφορά όλε τι αγορέ κάτω από 5 εκατομμύρια ευρώ. Και ο όρος θα πρέπει να πληρούνται ούτως ώστε κάθε φορά ε, να ισχύει το άρθρο 6 για την απόρριψη της προσφοράς. Ε, είναι όροι που επιβάλλονται αυστηρά, δηλαδή πρόκειται για μια περίπτωση που αφορά ένα αποθεματικό, ε, μια επιφύλαξη δηλαδή, σε σχέση με κάποια χώρα εταίρα, η οποία όμως αυτή η χώρα θα έχει υπόψη της ε, αυτή την επιφύλαξη, οπότε θα έχουμε την απόρριψη της προσφοράς για το ΑΒ προϊόν ή θα πρόκειται για κάποιο είδους δοκιμή πραγματικότητας όσον αφορά την ε, ουσιαστική αμοιβιότητα και όχι μόνο δηλαδή όσον αφορά το γράμμα και το κείμενο αλλά σε, βάση πρακτικής δραματικότητα. Και γι' αυτό το λόγο μέσα σε αυτό το σύστημα έχουμε και, την, και ένα επιπλέον επίπεδο ασφαλείας όσον αφορά την αγορά, ούτως ώστε ε, εάν συντρέχουν αυτές οι προϋποθέσεις να απορρίπτεται αυτή η προσφορά και είναι κάτι επομένω το οποίο θα ισχύει ε, από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία βλέπει αν πληρούνται οι όροι και προποθέσει. Οπότε έτσι να είναι δυνατόν να ενεργοποιηθεί αυτή η ε, δυνατότητα, αν θέλουμε να έχουμε ε, μια ελάχιστη μόχλευση για τις ε, διαπραγματεύσεις θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με το άρθρο 6 σε σχέση με το άρθρο 8 και το άρθρο 10 γιατί συχνά μέσω αυτών των κοινοποιήσεων δυνάμει του άρθρου 6 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να διαμορφώσει μια, μια ιδέα να έχει μια ιδέα για το τι γίνεται οπότε τότε ε, και ενεργοποιείται αυτού του είδους ε, η διάταξη, το άρθρο 8 ή το άρθρο 10. Οπότε έχουμε έτσι μια σφαιρική αντίληψη και άρα θα πρέπει να δούμε αυτά τα άρθρα, το ένα συνδυασμό με το άλλο, αν θέλουμε να, να έχουμε μια ολοκληρωμένη άποψη για την ρυθμίση αυτή. Είναι σημαντικό. Επίσης, ε, ο Επίτροπος ε, Μπαρνιέ αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα της λειτουργίας διότι οι υπηρεσίες αυτές ε, ε, ενέχονται άμεσα σε αυτές τις ε, διαπραγματεύσεις όσον αφορά την αναθεώρηση της συμφωνίας για τις δημοσίες συμβάσεις, οπότε και θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι είναι απαραίτητο να δούμε πώς θα είμαστε αυθεντικός διαπραγματευτής και να λαμβάνετε υπόψη ότι de facto υπάρχει άνοιγμα αυτών των αγορών των συμβάσεων και ο συνομιλητής να θεωρεί ότι είναι δεδομένο και εκτιμένο το ότι η προσβασιμότητα στην ε, ε, ευρωπαϊκή αγορά είναι δεδομένο. Μα τότε αν το θεωρεί αυτό τότε έχει λιγότερο ενδιαφέρον ή συμφέρον να, να, να μπει σε μια τέτοια σύμβαση, ένα τέτοιο διαγωνισμό η προμήθεια. Οπότε η Ευρώπη αφού θέλουμε να έχει τέτοιου είδους ε, πρόσβαση στις αγορές των χωρών, τότε θα πρέπει να προσφέρει αντιστάθμισμα κάπου, κάπως. Και θα πρέπει σε κάποια, σε κάποια άλλη, άλλη, άλλη διάσταση, άλλη πτυχή της ελεύθερης συναλλαγής να προσφέρει το αντιστάθμισμα. Επομένως, ξέρουν εκείνοι ότι είναι ανοιχτή η αγορά. Τότε ανοίγουν ή δεν ανοίγουν ε, την δική τους αγορά. Ξέρουν, επομένως, ότι εμείς έχουμε τη δική μας αγορά ανοιχτή Οπότε τότε προσπαθούν να δουν πώς θα, θα αποσπάσουν κάτι, γιατί ξέρουν ότι αν θέλουμε να, να μπούμε στην αγορά τους, κάτι πρέπει να δώσουμε αλλού. Ναι, γι' αυτό σας λέω ότι υπάρχει εδώ αυτή η ευαισθησία, αυτή, αυτό το λεπτό σημείο, το οποίο νομίζω ότι το έχει πει ο κύριος ε, Μπαρνιέ. Είναι κάτι δηλαδή πάνω από την οδηγία, πέρα από την οδηγία, αλλά έχει σχέση με το θέμα μας, τις ε, δημόσιες συμβάσεις. Τότε θα πρέπει επομένω να έχουμε υπόψη μας ότι πρέπει να αναπτύξουμε αυτή την πτυχή του θέματος, αυτό, αυτή την, την, την, την μόχλευση. Πρόεδρος, σας παρακαλώ απαντήστε την ερώτησή μου. Δηλαδή σε σχέση με την εφαρμογή των ισχυρουσών διατάξεων όσον αφορά ε, την ε, οδηγία για τις ε, δημόσιες συμβάσεις. Τι γίνεται, ποιοι επικαλούνται αυτή την οδηγία είναι σημαντικό. σωστά; Και απαντήστε και αυτό που είπε η συνάδελφος. Γιατί είπατε ότι δεν έχουμε αρκετά στοιχεία. Τι, τι, τι, λέτε για αυτή τη ε, μελέτη επιπτώσεων. Όσον αφορά τη μελέτη των επιπτώσεων, νομίζω ότι η Επίτροπη σε όλα μας τα, τα, τα έγγραφα και εν παραρτήματι έχουμε εκεί ε, αριθμητικά στοιχεία, ε, τα εξηγούμε όλα, ιδίω όσον αφορά τα παρατήματα για να μην μπερδεύεται ο χρήστη ο αναγνώστης. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί τη βάση των διαθέσιμων στοιχείων ε, αξιοποίησε όσο μπορούσε περισσότερο αυτά τα στοιχεία υπολογισμού επί τη βάση κάποιων υποθέσεων. Και αυτές οι υποθέσεις ε, έχουν ενταχθεί στο κείμενο. Σε αυτή την θεματική είναι όταν δεν έχουμε δεδομένα για παράδειγμα για τα άρθρα 58 και 59 της ε, οδηγίας για αυτούς τους κλάδους και το πρόβλημα ότι δεν έχουμε κανένα είδους επιστροφή όσον αφορά την πραγματική λειτουργία γιατί ε, από καιρού καιρών ε, έχουμε κάποιο, κάποιο αίτημα, κάποιος ρωτά πώς μπορούμε να επικαλεστούμε, να αξιοποιήσουμε αυτές τις διατάξεις και υπάρχουν κάποιες ενδείξεις για το τι μπορούμε να κάνουμε. Δεν έχουμε επομένω κάποιο είδους αριθμητικά στοιχεία για να δούμε πώς θα μπορούμε να, αξιο, να αξιοπλογήσουμε ε, την, ε, την κατάσταση. Αλλά όμως είναι αυτή η μόνη, ε, η μόνη νομική βάση ούτω ώστε να μπορεί αυτός ο οποίος κάνει το διαγωνισμό να απορρίψει μια προσφορά. Οπότε γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να βλέπουμε κάθε φορά εάν έχει τα στοιχεία που χρειάζονται γιατί ε, σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται να υπάρχει μια συγκεκριμενοποίηση για το πώς μπορούν τα στοιχεία να χρησιμοποιηθούν. Και για αυτό και έχουμε εντάξει στην μελέτη των επιπτώσεων όλα τα στοιχεία τα οποία έχουμε στη θέση μας. Αλλά επίσης ξέρουμε σε ποια σημεία δεν έχουμε στοιχεία και έτσι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε και να συγκεκριμενοποιήσουμε την αξιολόγηση. Και εγώ θα ήθελα να προσθέσω κάτι σύντομο όσον αφορά τη μέρη των επιπτώσεων. Γιατί ε, υπάρχει εδώ μια παρεξήγηση. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όταν κάνουμε των επιπτώσεων, έχουμε δύο, ε, δύο, δύο, δύο, φορές εξετάζουμε ε, το, το, το, θέμα. Γι' αυτό και την τελευταία φορά είχαμε ε, κάποια ζητήματα που ανέκυψαν που επιδεχόντο ε, βελτίωση. Οπότε έχουμε την τελική μορφή, την τελική αξιολόγηση, όπου αξιολογούμε τα πάντα, όλα τα δεδομένα. Όμως αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε με τους ισχύοντες κανόνες είναι να κάνουμε ε, μία τρίτη εξέταση, ούτω ώστε να μπορούμε να επικυρώσουμε κατά κάποιο τρόπο ε, τα, τα προηγούμενα στοιχεία. Άρα, επομένως, αυτό που θα να κάνουμε και το έχει στο Ιντερνετ, να, να καλύψουμε τα, ό,τι μας απασχολεί για να, για να δούμε τη δεύτερη και οριστική γνωμοδότηση και αξιολόγηση. Δεν μπορούμε να το κάνουμε όμως για τρίτη φορά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η τελική μορφή. είναι ό,τι τροποποιήθηκε αφού λάβαμε από την Επιτροπή που εξετάζει τα, τα, τα σχόλιά της. Και τώρα κάτι άλλο, σε αυτό το τελευταίο παράρτημα, για την μελέτη των επιπτώσεων, ακριβώς εκεί αναφέρει σε ποιο σημείο και με ποιο βαθμό η Επιτροπή, οι υπηρεσίε μας δηλαδή προσπάθησαν να καλύψουν, να λάβουν υπόψη ε, τα, τα αιτήματα της Επιτροπής της αξιολόγησης των επιπτώσεων. Και εκεί μπορεί να δείτε πώς επεξεργαστήκαμε ή επανεπεξεργαστήκαμε την ε, αξιολόγηση των επιπτώσεων. Προεκτικομένως για ένα έγγραφο εργασίας. Οπότε ε, εμείς αποφαινόμεθα επί τη βάση αυτών των εγγράφων, αλλά έχουμε και την τελική λέξη, την τελευταία λέξη, σε σχέση με το αν υπάρχει κρίσιμη μάζα ούτως υπήν των, ε, των ε, πληροφοριών. Κατά κάποιο τρόπο είναι πολιτική απόφαση, το τι να αντιθούν αυτά υπόψη και να υπάρχουν τα, τα δεδομένα, ε, τα διαθέσιμα, ούτως ώστε να αποφασίσει η Επιτροπή κατά πόσον θα προχωρήσει σε κάποιο πρόγραμμα ή όχι. Έρχεται επομένως ε, αυτό να συμπληρώσει το έγγραφο που υπάρχει, το οποίο όμω ποτέ δεν μπορεί να είναι τέλειο, γιατί ποτέ δεν έχουμε όλα μα όλα τα δεδομένα. Πρόεδρο. Η οχι ερχεται επομένω. αυτο να συμπληρωσει το εγγραφο που Βάιλερ, πρώτα πρώτα. Σας ευχαριστώ για τις τόσο πλήρες απαντήσει σα. Έχουμε, έχουμε χρόνο. Οπότε μπορούμε να έχουμε και κάποιες ερώτα-απαντήσεις Κυρία Βάιλερ, εσείς είχατε ζητήσει πρώτο λόγο, αν θυμάμαι καλά. Και κατόπιν, ε, λέω και κατόπιν ο κύριος Σουβάμπ θέλει να επανέλθει ως εισηγητής. Ευχαριστώ. <clears throat> Για τα GPS εξήγησατε, γιατί δεν είναι συγκρίσιμη κατάσταση με αυτό εδώ το νομοθέτημα. Όμω δεν απαντήσατε στη δική μου ερώτηση. Γιατί δεν φροντίζουμε σε σχέση με, τους πιο, με τον πιο ισχυρό, τον πιο μεγάλο ε, εμπορικό μας εταίρο, τι ΗΠΑ, να αποφασίσουμε τι θέλουμε. Γιατί χρειάζεται αυτή, αυτό το νομοθέτημα εφόσον φτιάχνουμε ε, Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών και ξέρουμε ότι στις δημόσιες προμήθειες, εξοπλισμούς και υψηλής τεχνολογικής ε, αξίας προϊόντα δεν έχουν ανοιχτέ τις αγορές τους Αμερικανοί. Ίσως λοιπόν θα μπορούσαμε να βρούμε τη λύση χάρη στην ε, Συμφωνία των Ελεύθερων Συναλλαγών. Και κάτι άλλο. Και το υπογραμμίσω. Είπατε ότι είναι πολύ οικονόμα τα κράτη στην Ευρώπη στις δημόσιες προμήθειες. Δηλαδή πρέπει να δώσουμε ευκαιρίες ε, στις εταιρείες της Ευρώπης να ανοίξουν δρόμους που δεν είχαν μέχρι τώρα. Ναι, είναι κάτι που συζητούμε και σε εθνικό επίπεδο. Αλλά εμείς θα προτείναμε σαν λύση να πείσουμε εν τέλει τα δημόσια, τα κρατικά, τις κρατικές αρχές να επενδύουν στις υποδομές. Αλλά είναι ενδιαφέρον αυτό που λέτε είναι κατεπήγον να αρχίσει να επενδύει, και αυτό το ισχύει ξεκάθαρα και συζητείται ήδη στη Γερμανία, το κράτος, ε, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να αλλάξει πολύ γρήγορα. Ευχαριστούμε πολύ για τις απαντήσεις που μας δώσατε. Για να είμαι σαφής ε, στο ερώτημα σχετικά με τα ευρήματα, είπατε πολλά και τα αποδεικτικά. Ε, είπατε πολλά και σέβομαι τα βασικά σας στοιχεία. Απ' την άλλη πλευρά, έτσι όπως τα καταλαβαίνω αυτό που μας είπατε, είναι ότι εάν δεν έχουμε τα στοιχεία για να υλοποιηθούν, ε, μάλλον για να... Ε, γίνουν ε, τα ευρήματα πιο σωστά, ε, χρειάζονται περισσότερα στοιχεία. Δηλαδή δεν έχετε ακριβώς ε, όλα τα στοιχεία που χρειάζεστε. Νεύετε αρνητικά, σημαίνει ότι δεν κατάλαβα καλά. Εντάξει. Αναφερθήκατε στο άρθρο 6 και είπαμε ότι υπάρχουν δύο επικαλυπτόμενες διαδικασίες δεν είναι, ε, αληθεύει ότι αν χρησιμοποιήσουμε τα άρθρα 6 και τα άρθρα 8 μέχρι 10 ή 11 ε, τότε θα ε, διακινδυνεύουμε δύο επικαλυπτόμενες διαδικασίες. Σας ευχαριστώ πολύ και κάτι άλλο από μένα, εάν μου δίνετε την άδεια να ρωτήσω. Είναι κάτι που ρώτησε η κυρία εαν μου δινετε την αδεια να ρωτησω ειναι κατι που ρωτησε η κυριε βαιλερ Ο κύριος Γέντσεν είναι από ό,τι φαίνεται ε, έμπειρος, πολύπειρος ε, διαπραγματευτής εμπορικός ξεκινάνε σε λίγο ε, οι εμπορικές συμφωνίες δεν θα, λέτε, δεν θα ανοίξουν εάν δεν συμφωνήσουμε από αυτό. Μα δεν θα υπάρξει συμφωνία πριν από 5-6 μήνες. Νομίζω ότι η θέση είναι, λέμε, ότι μία από τις αρχές της Ευρώπης είναι ότι είμαστε ανοιχτοί και αυτή είναι η ισχυρή μα θέση στι διαπραγματεύσεις, στις εμπορικέ διαπραγματεύσεις. Όμως τώρα αποφασίσαμε με τα κράτη-μέλη ότι θα βάλουμε και κάποιους κανόνες ε, έτσι ώστε να αλλάξουμε την κατάσταση αν δεν μας δώσετε αυτά που ζητάμε. Έτσι είναι. Ευχαριστώ. Να επανέλθω. Γιατί χρειαζόμαστε λοιπόν αυτή τη συμφωνία με τις ΗΠΑ. Ε? ή με άλλον. Προσπαθούμε να αλλάξουμε νοοτροπίες. Το σύστημα πρακτικά λειτουργεί ως εξής. Ξεκινάνε διαπραγματεύσεις με ε, τις ομάδες των εμπειρογνωμόνων, ας πούμε, τις ομάδες μας και των άλλων κρατών που είναι υπεύθυνε ε, για δημόσιες συμβάσεις. Ε, δεν μπορούμε να τους πούμε όλα τα μεμονωμένα προβλήματα που έχουν ε, οι εταιρείε μας. Ε, συνήθως είναι πολύ ευγενεί, χαμογελούν ναι. ευγενικά, αλλά δεν πολύ έχουν διάθεση να συζητήσουν σε λεπτομέρεια τις δημόσιες συμβάσεις. Κυρίως σε επίπεδο δημόσιων ε, συμβάσεων σε επίπεδο ομοσπόνδων ε, κρατών, σε επίπεδο πολιτιών δηλαδή, στις ΗΠΑ η πρόσβαση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Στις ε, εμπορικές διαπραγματεύσεις κάτι παίρνεις, κάτι δίνεις. Επομένως δεν καταλαβαίνω εδώ γιατί πρέπει να πληρώσω ας πούμε για κάτι το οποίο ήδη μου δίνει. Είναι λίγο αυτή η υπεραπλουστευμένη μένα, αλλά αυτή είναι η σκέψη των εμπορικών εταίρων. Αυτό στην ουσία σημαίνει και νομίζω ότι ο συνάδελφος το έθιξε αυτό προηγουμένως. Θέλουν ε, δεσμεύσεις αλλού λένε ωραία θέλετε καλύτερα πρόσβαση για τις επιχειρήσεις σας, ωραία το καταλαβαίνουμε. Αλλά εάν το θέλετε αυτό θέλουμε να κάνετε υποχωρήσεις ε, και να μας παραχωρήσετε πράγματα σε, άλλες, ε, σε άλλους χώρους. Δεν θέλουν να πολυσυζητήσουν, δεν θέλουν να παίξουν με τις δημόσιες συμβάσεις γιατί δεν πιέζονται από τις εταιρείε τους γι' αυτό. Θέλετε πρόσβαση, ωραία, αλλά και εγώ πρέπει να είμαι σε θέση να δώσω στους ψηφοφόρους μου κάτι σε αντάλλαγμα. Και επομένως αυτή είναι, αυτό είναι το πνεύμα μέσα στο οποίο ξεκινούν ε, οι συζητήσεις. Και επομένως γι' αυτό λέω ότι τέτοια ε, συζήτηση Δηλαδή, ναι, εντάξει, στην ουσία μας λένε, αν θέλετε ναι, μπορούμε να το συζητήσουμε, αν θέλετε ναι, μπορούμε να ε, ε, ε, διασφαλίσουμε κάποια πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις, αλλά μην νομίζετε ότι θα είναι για πάντα και για όλη τη ζωή. Επίσης, είναι πολλές και διαφορετικές οι απόψεις τις οποίες έχουμε απέναντί μας. και ούτε μπορούμε να πούμε κλείνουμε τις αγορές και μετά τις ανοίγουμε σιγά σιγά και καταδοδοκούν. Όσον αφορά τα δεδομένα, δεν είπα ότι δεν έχουμε δεδομένα αυτό που αναγνωρίζουμε είναι ότι τα στοιχεία για τις δημόσιες συμβάσεις είναι ατελή αυτή τη στιγμή για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και για προηγμένες οικονομίες Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και Ηνωμένων Πολιτειών. Έχουμε διαφωνίες όσον αφορά τα στοιχεία, τα δεδομένα. Εάν δεν ξεφύγουμε από τις Ηνωμένε Πολιτείες, τότε οι διαστάσεις είναι πολύ μεγάλες. Ε, οι αριθμοί δεν ταυτίζονται. Φανταστείτε τι γίνεται με τις κινέζικες δημόσιες ε, συμβάσεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε με τη μελέτη αντικτύπου αναγκαστήκαμε να ξεκινήσουμε και από κάποιες ε, ε, αρχές και κάποιες ε, υποθέσεις εργασίας και βεβαίως παραδεχόμαστε ότι δεν είναι το τέλειο προϊόν γιατί δεν μπορούμε να έχουμε στοιχεία για όλα τα πράγματα. Αυτό είναι ένα εργαλείο το οποίο δημιουργήθηκε για να βοηθηθούν οι πολιτικοί υπεύθυνοι όταν θα πάρουν κάποιες αποφάσεις, αλλά ακόμα δεν έχουμε τα τέλεια στοιχεία για την ώρα κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε με αυτές τις ελλειπείς πληροφορίες, κυρίως δε όταν αναφερόμαστε για το πλαίσιο εκτός Ευρώπης. Δεν, βρισκό, δεν βλέπουμε αντίφαση. Εμείς προσπαθούμε απλώς να αλλάξουμε λίγο την οτροπία των ε, ε, εταίρων, να αλλάξουμε λίγο τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται, να πούμε να έχουμε μια ανοιχτή αγορά, αλλά ξέρετε να είστε σοβαροί όταν σας μιλάμε για δημόσιες συμβάσεις, ε, δηλαδή ε, ναι, εμείς είμαστε ανοιχτοί, αλλά και εσείς πρέπει να κάνετε κάτι. Ε, και εσείς πρέπει να μας δώσετε κάτι. Στην ουσία δεν μπορεί κανείς να πληρώσει για να έχει ε, ανοιχτή αγορά. Θα έπρεπε να είναι συνειφασμένο με την ίδια την αρχή των δημοσίων συμβάσεων. Όσον αφορά τώρα το ζήτημα το οποίο σχετίζεται με τις ε, παράλληλες διαδικασίες ε, άρθρο 6 και άρθρο 8 μέχρι 10 και τις ενδεχόμενες επικαλύψεις που αναφέρατε. Είναι γεγονός ότι de facto μπορεί να βρεθούμε σε κατάσταση όπου μπορεί να έχουμε την ε, απόφαση μιας αρχής η οποία αποφαίνεται επί της συμβάσεων και η Κομισιόν να πρέπει να δώσει την άποψή της, αλλά αυτό σημαίνει η Κομισιόν όμως ε, ε, βάσει των ευρημάτων, βάσει των στοιχείων που έχει στη διάθεσή της ε, διαπιστώνει ότι είναι λίγο αρρωστημένη η κατάσταση, είναι ασθενή λίγο ο τομέας αυτός. Στα πλαίσια της ε, μεμονωμένης ε, κοινοποίησης ε, βρίσκει εφαρμογή στο άρθρο 6 όμως, υπάρχουν και τα άρθρα 8 με 10, τα οποία προβλέπουν ένα πιο ευρύ πλαίσιο πέρα από τη, τις συγκεκριμένε περιπτώσεις διότι μίλης ότι αντίθετα από το άρθρο 6 το, τα άρθρα 8 με 10 έχουν μεγαλύτερο εύρος και έχουν μεγαλύτερο πεδίο εφαρμογής από ότι το άρθρο 6 η συνοχή πρέπει να υπάρχει και πρέπει να μείνει μέχρι το τέλος της διαδικασίας. Και κατά αυτό το πνεύμα έχουμε κάνει αυτές τις προτάσεις. Αλλά βεβαίως πάντοτε θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε κάθε πρόταση που μπορεί να έρθει στη διάρκεια της ε, διαπραγμάτευσης και που μπορεί να προτείνει κάποια βελτίωση. Όμως επί της ουσίας ε, για τον τρόπο με τον οποίο όπως σας εξήγησα διαρθρώνονται οι δύο διαδικασίες δεν υπάρχει πρόβλημα ε, και δεν υπάρχει είτε ασυνέπεια είτε ασυνέχεια. Να... Αν μου επιτρέπετε να και εγώ κάτι. Σε ένα επιπλέον εγγύηση ότι δεν θα διαταραχθεί τίποτα από τις διαδικασίες. Το άρθρο 9 και παράγραφος 4 προβλέπει ανασταλτική ανασταλτικό αποτέλεσμα από τη στιγμή που ένα κράτος δηλώνει ότι είναι να να ε, ξεκινήσει διαπραγματεύσει. Από εκεί και πέρα δεν γίνεται δυνατή η επίκληση του άρθρου 6 και νομίζω ότι σε αυτό το παράδειγμα αναφέρεστε. Απάξ και αρχίσουμε δηλαδή μαζί με ένα τρίτο κράτο να ε, διαπραγματεύσουμε, να διαπραγματευτούμε. Δεν μπορεί ε, ένα κράτος μέλος, Φερρυπίνη, οι αρχές αρχή της Δανίας που αναφέρατε, να ζητήσουν την εφαρμογή, την ενεργοποίηση του άρθρου 6. ο Πρόεδρος. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Σας ευχαριστώ όμως και πρέπει να σταματήσουμε. Δίνω το λόγο στον κύριο Σφάπ ως αναπληρωτή εισηγητή ή συντάκτη για να μας ε, πει. Ευχαριστώ πολύ, πολύ Πρόεδρε. Να σας πω και να σχολιάσω με όλο το σεβασμό προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κοιτάξτε, ε, υπάρχουν πολλέ φορέ σκέψει για το θέμα αυτό. Αλλά νομίζω ότι κάπω το, το, το έχουν παρακάνει τώρα. Γιατί προσπάθησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συγκεράσει αυτέ τι ε, σχολέ σκέψει. Και ε, δεν ξέρω, είναι πάρα πολύ δύσκολο τώρα να, να, να, να το τι γίνεται. Νομίζω ότι δεν υπάρχει ισορροπία. Δεν είναι καλά σταθμισμένα τα όσα λέει η Επιτροπή, κάποιοι φίλοι από τις νότιες χώρες δεν είναι εδώ. Να σας πω τι, έγινε πέρσι. Στο Βερολίνο είχαμε συζητήσει με συναδέλφους ε, από το κόμμα μας και ήταν και κάτι σύμβουλοι κάποιων εταιριών. Οπότε ε, υπήρχε κάποιο μόνο πάρα πολύ έμπρο και αυτό είχε πει όταν τον ρωτήσαμε ότι χρειάζεται περισσότερη αμοιβαιότητα. Αυτό ε, ενεργοποιείται στον, ε, δραστηριοποιείται στον, ε, στο χώρο του γυαλιού. Για τις εξαγωγές, επομένω, δεν επιθυμητά αυτό το οποίο προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επίσης ε, έχουμε και κάποια εταιρεία γαλλική για είδη πολυτελείας οι οποίοι λέγανε ότι όχι μην κάνετε κάτι αυτό που προτείνετε γιατί τότε θα βάλετε εν κινδύνο όλες με τις εξαγωγές. Είδατε. Η κάθε σχολή έχει ε, άλλη σχολή σκέψης λέμε αλλά δεν είναι αλήθεια. Και ένας μεγάλος παραγωγός λοιπόν γελιού που ήθελαν περισσότερη αμοιβιότητα αυτοί παράγουν το αλλά άλλο κομμάτι της, ε, της εταιρεία έλεγε όχι, ε, μην, το κάνετε αυτό, θα χάσουμε την αγορά. Άρα τελικά όλα εξαρτώνται από το για ποιο κομμάτι της αγοράς, για ποιο κλάδο ακριβώς μιλάμε. Μιλούμε επομένως εδώ για τις αγορές που αφορούν τις ε, συμβάσεις αυτές. Δηλαδή είναι ευρύτερο το θέμα. Τώρα, σε σχέση με αυτό που είπε η κυρία Βάιλερ, ισχύει το ότι αυτού ε, του γενικευμένε προτιμήσει, εάν γίνει συμφωνία με την Ιαπωνία, που είναι λίγο αισιόδοξο, τότε θα έχουμε και άλλες χώρες, όπως ο Καναδάς. Και αυτό το GPA, τη Συμφωνία Γενικευμένων Προτιμήσεων, δεν έχει υπογράψει. Καναδάς και άλλες χώρες. Και μας είπε ο Καναδάς ότι υπάρχει εδώ στοιχείο βιότητας. Δεν έχουν συμφωνήσει όλε τι χώρε με αυτό, ότι θα πρέπει να είναι οι αγορέ ανοιχτέ. Μόνο οι μισέ είναι ανοιχτέ, όπω είπε η κυρία Ρίλε. Άρα, επ' αυτού θα πρέπει να προσέξουμε πώ θα ανοίξουμε όλε τι αγορέ. Δεν έχω πιστεί ότι βρέθηκε η λύση. και είναι δικαιολογημένε όλε οι επικρίσει κατά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη πρότασή τη. Θα το ξανασυζητήσουμε στην Επιτροπή μα και στην Επιτροπή Διεθνού Εμπορίου. Οπότε θα διαπιστωθεί ότι η μέση οδός είναι η πιο σωστή και από αυτού αποφασίσει το Κοινοβούλιο. Σα ευχαριστώ πολύ. Το ερώτημα είναι αν μπορεί να βρεθεί κάποια λύση εδώ ή κάποια δυνατότητα. Ο κύριος Έγγελ θα στείλει τη γνωμοδότησή του στη μετάφραση στις αρχές Μαΐου. Στις, ε, τον ε, Ιούνιο θα συζητήσουμε, 11 Ιουλίου είναι η, πρόθεση, η, συγγνώμη, η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών και Σεπτέμβριο στην Ολομέλεια. Στις 25-26 Σεπτεμβρίου όμως λέμε ότι θα συζητηθούν ε, οι αντιφατικές ε, ε, τροπολογίες, άρα αργότερα θα πάμε στην Ολομέλεια. Ναι, ναι, έχετε δίκιο. Έχουμε μέχρι το Σεπτέμβριο λοιπόν. και στις 27, 26, 27 Νοεμβρίου θα ψηφιστεί το θέμα στην Επιτροπή Εξωτερικού Εμπορίου. Διεθνούς μάλλον εμπορίου. Πάρα πολύ ωραία. Ε, Σα ευχαριστώ όλους. Μπορούμε να περάσουμε τώρα στο επόμενο θέμα. Είναι δικιά μου γνωμοδότηση. Κράτησε λίγο παραπάνω το προηγούμενο θέμα και επομένως ε, μας περιμένει και η Κομισιόν για το θέμα αυτό που είναι εδώ και ο κύριος Σμίτ είναι εδώ ναι, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Σας καλωσορίζουμε και συγγνώμη που καθυστερήσαμε λίγο και περιμένατε. Χαίρομαι λοιπόν που μπορώ να παρουσιάσω την πρότασή μου. Ο κύριος Κάμπος είναι εδώ, δεν βλέπω. Ε, ο κύριος Μάντος δεν είναι εδώ. Α, ο κύριος Σμίτ προσωπεί τον κύριο Μάντας, πάρα πολύ. Η κυρία Ρούλε είναι εδώ, αλλά δεν ξέρω, είναι σκιώδης συγγετρία, είστε. Α. Καλωσορίσατε, λοιπόν και για αυτό το θέμα. Μήπως θα με προσέχατε λίγο, λέει ο Πρόεδρος. Την προσοχή της κυρίας Ρούλε ήθελα, αλλά... From the uh, Commission is a new regulation EU rules um, rules across the European Union on Λοιπόν, περιοδικός τεχνικός έλεγχος των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρημουλκούμενών τους. Ευαίσθητο θέμα το οποίο αφορά και την προστασία των καταναλωτών και την προστασία βεβαίως του περιβάλλοντος γνωρίζετε ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τον, την προσέγγιση ε, και την αντιμετώπιση αυτών των περιοδικών, τακτικών, τεχνικών ελέγχων. Είτε πρόκειται ε, για την περίοδο μεταξύ των τεχνικών ελέγχων, είτε ε, πρόκειται για το ίδιο το περιεχόμενο του τεχνικού ελέγχου, ο τύπος των μηχανοκινήτων οχημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής, καθώς επίσης μερικές φορές και ίδια η η ποιότητα και η προσοχή που δίνεται στην διασφάλιση της ποιότητας κατά τη διάρκεια αυτών των τεχνικών ελέγχων. Όλα αυτά τα στοιχεία από πλευρά της δικής μας Επιτροπής ε, φαίνεται να αποτελούν ε, ε, κατά κάποιο τρόπο αρμοδιότητα της Επιτροπής Μεταφορών. Σε όρους ενιαίας αγοράς δεν υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να γίνονται οι τεχνικοί ε, έλεγχοι. Έκανα και κάποιες ε, προτάσεις κατά αυτήν την έννοια και σχετικά και με την ε, μετακίνηση των οχημάτων ε, και ο κύριος ε, Μάντερς θα συνεργαστεί και συνεργάζεται ήδη μαζί μου γιατί βλέπει το θέμα από την πλευρά της οδηγίας για την ταξινόμηση των οχημάτων. Στην ουσία εδώ μιλάμε και για την αμοιβαία αναγνώριση των τεχνικών ελέγχων ασφαλείας γιατί αυτό είναι ένα από τα κυριότερα, κεντρικότερα σημεία και στοιχεία της πρότασης της Κομισιόν. Ε, θα κάνω κάποιες ε, ε, προτάσεις, τις οποίες γνωρίζω ότι θα ακούσει έτσι με συμπάθεια η Κομισιόν. Γιατί ξέρω ποια είναι και η θέση τους για την έννοια αγορά. Όσον αφορά τις ε, χώρες ας πούμε οι οποίες ε, είναι κύρια αναμειγμένες ε, και στο ζήτημα της μεταφοράς ταξινόμησης. Η χώρα στην οποία μεταφέρθηκε το αυτοκίνητο ε, και ε, ε, την εποχή που είχε ας πούμε δύο χρόνια ακόμα μπροστά του μέχρι να γίνει ο επόμενος τεχνικός έλεγχος και αν πήγε στη διάρκεια της πρώτης χρονιάς ισχύω του πιστοποιητικού τεχνικού ελέγχου στην ελόγω χώρα αυτό σημαίνει ότι τον επόμενο χρόνο θα πρέπει να κάνει ένα νέο τεχνικό έλεγχο. Επίσης σε μερικές περιπτώσεις λέμε ότι κοστίζει περισσότερο ο τεχνικός έλεγχος από ό,τι σε άλλες χώρες. Εγώ δεν είμαι σίγουρη σίγουρος ότι αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα. Το σημαντικό είναι να έχουμε ε, ε, ε, τεχνικούς ελέγχους, ε, ελέγχους ποιότητας που να είναι υψηλού επίπεδου, ταυτόσιμου επίπεδου παντού. Όσον αφορά τις τροπολογίες που έχω υποβάλει, να σας πω ότι προσπάθεια να ε, προσθέσω ε, αξία υπό το φως των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής ΙΜΚΟ Πρέπει να δούμε λοιπόν την ε, διασύνδεση του περιοδικού τεχνικού ελέγχου ε, σε σχέση να, δούμε τη διασύνδεση μεταξύ αυτής της οδηγίας και της ε, οδηγίας που ασχολείται με τα τεχνικά ζητήματα των αυτοκινήτων που διακινούνται προς πώληση γενικά. Στα παραρτήματα βεβαίως υπάρχουν και πάρα πολλές τεχνικές λεπτομέρειες, αλλά πρέπει να σας πω ότι είναι σαφές και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ένα νέο όχημα ε, με τα χρόνια μπορεί να τροποποιηθεί. Πρέπει κανείς ε, να είναι πάρα πολύ προσεκτικός έτσι ώστε να παραμένει λογική και σωστά διασυνδεδεμένη με τις άλλες οδηγίες αυτή η οδηγία. Και επίσης ε, ο περιδιωκός τεχνικός έλεγχος θα πρέπει να γίνει με βάση τα στοιχεία τα οποία θα έπρεπε να έχει το όχημα από την αρχή της ζωής του, από τη στιγμή της πρώτης του πώλησης. Ε, κάνω κάποιες ε, τροπολογίες λοιπόν γι' αυτό για να αποσαφινιστούν κάποια πράγματα. Δεύτερο σημείο, το θέμα της προστασίας ε, των καταναλωτών. Γιατί αν δει κανεί ε, το scoreboard, τον πίνακα επιδόσεων της εσωτερικής αγαράς, διαπιστώνει ότι ο τομέα τη αγορά που έχει μικρότερο ποσοστό ικανοποίηση καταναλωτών και μάλιστα είναι η τρίτη συνεχής χρονιά με το ίδιο αποτέλεσμα, είναι ο τομέας των οχημάτων. Βεβαίως εδώ δεν μπορούμε να λύσουμε ή να αντιμετωπίσουμε όλα τα προβλήματα τα οποία αφορούν ε, την, ε, ε, τα, αυτοκίνητα από δεύτερο χέρι, την παρουσία τους, τον τεχνικό τους έλεγχο, το ένα το άλλο. αλλά το ζήτημα είναι να μπορούμε να αποφύγουμε τις απάτες και τις επισκοπού εσφαλμένες πληροφορίες. Ε, κυρίως όσον αφορά το, ε, τα χιλιόμετρα, το κοντέρ. Ε, ξέρουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις το κοντέρ είναι πειραγμένο όταν φτάνει το αυτοκίνητο να πολιθεί και επομένως θα πρέπει να υπάρχει κάποια πρόνοια η οποία να μπει σε αυτήν την οδηγία η οποία να προβλέπει κάποια τροποποίηση της ε, κατάστασης. Ένα άλλο ε, σημείο το οποίο γνωρίζουν πολύ καλά, το έχουν δουλέψει οι βουλευτές αυτής ε, της Επιτροπής, είναι η πρόσβαση σε τεχνικές πληροφορίες έτσι ώστε να ελέγχονται τα οχήματα, ας πούμε, για, την, για τα, σύστημα πέδησης, για τα συστήματα πέδησης ή για, τα, για τις εκπομπές αερίων κτλ. είχαμε και μία άλλη έκθεση για το Euro 6 που ε, είχε μεγάλη σημασία δώσει σε, αυτήν, την, σε αυτόν τον έλεγχο ε, και στην συμβατότητα των ε, ε, ελέγχων, συγγνώμη, των κέντρων τεχνικού ε, ελέγχου ε, και αναφερόταν τότε ότι σε μερικέ περιπτώσεις ο τεχνικός έλεγχος γίνεται από πάρα πολύ μεγάλα γκαράζ, από γκαράζ που δεν είναι ανεξάρτητα, ενώ στη δικιά μου χώρα γίνονται οι έλεγχοι αυτοί από, ανεξάρτητες, από ανεξάρτητα συνεργεία, τα οποία μάλιστα είναι και πάρα πολύ προσεκτικά. και να σας πω ότι έχω και ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι έτσι η αντίκα και το οποίο έχει πάρα πολύ λίγα χιλιόμετρα ε, και ήρθαν τόπου οι ελεκτές για να δουν αν πραγματικά στη διάρκεια του τεχνικού ελέγχου αν πραγματικά ήταν έτσι και δεν είχα πειράξει το κοντέρ. και μάλιστα στην πρώτη συζήτηση τότε είχε αναφερθεί ότι δεν είναι δυνατόν να γίνονται τέτοιου είδους έλεγχοι από το Ηνωμένο Βασίλειο ε, και εγώ είπα ότι εμείς πάντα τους κάναμε τους ελέγχους αυτούς και επομένως ε, δεν είναι δυνατόν να μην τους κάνουμε. Λοιπόν, ε, θα πρέπει να διασφαλιστεί η παρουσία σωστών οργάνων στο σημείο που γίνεται ο τεχνικός έλεγχος ε, και κυρίως όταν πρέπει να ελέγξουν ήδη περίπλοκα μηχανήματα όπως είναι ας πούμε ε, τα γεωργικά μηχανήματα ή τα τρακτέρ. Ε, όσον αφορά τα συλλεκτικά αυτοκίνητα, ιστορικά αυτοκίνητα κτλ. Αντίκες. Εγώ έχω ένα αυτοκίνητο που είναι 24 χρόνων. Όταν θα γίνει 30 ε, χρόνων θα πρέπει να περάσει από γενικότερο τεχνικό έλεγχο. Αυτό το αυτοκίνητο κάνει περίπου 5.000 χιλιόμετρα το χρόνο ε, και το προσέχω πάρα πολύ. Δεν ε, ακολουθεί έτσι συνήθεις διαδικασίες κυκλοφορίας, αλλά παρόλα αυτά στα 30 θα πρέπει να περάσει ένα πολύ μεγάλο τεχνικό έλεγχο. Νομίζω ότι και ο καθορισμός των ε, συλλεκτικών αυτοκινήτων και των ε, αντικών θα πρέπει ε, να παραμείνει, να παραμείνει η δικαιοδοσία των κρατών μελών. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος εδώ πλήρως να περιγραφεί το τι εννοούμε με αυτοκίνητα αντί και συλλεκτικά. Επίσης έχω βάλει για κάποια άλλα στοιχεία όσον αφορά την αμοιβαία αναγνώριση. Υπάρχουν και κάποια σημεία τα οποία σίγουρα θα ξαναβρείτε στις ε, εκθέσεις της Επιτροπής ε, Μεταφορών. Ελπίζω ότι η Κομισιόν θα δει με συμπάθεια της, ε, την προσπάθειά μας. Ελπίζω ότι και οι σκιώδεις ηγητές θα καταλάβουν το πνεύμα των προτάσεων, αλλά βεβαίως, βεβαίως θα περιμένω και από τη δική τους πλευρά να δω κάποια συνεισφορά. Ε, με μεγάλη ευχαρίστηση λοιπόν θα ακούσω τα σχόλιά σας, αλλά ίσως πριν η Κομισιόν θέλει να μας πει δύο λόγια και να μας πει και πώς θα συνεχίσουμε, πώς θα προχωρήσουμε. Βάντεν Κάπ. Ε, Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Και ευχαριστώ για τη σαφή αυτή τοποθέτηση γνωμοδότηση. Έχει μια σαφή προοπτική ΙΜΚΟ. Στις κάτω χώρες το θέμα αυτό έχει μεγάλη πολιτική σημασία και πιστεύω ότι θα βοηθήσει και την εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η γνωμοδότησή σας. Γιατί μπορεί να μην γνωρίζει ο Ολλανδός τι είναι οι δημόσιες προμήθειες ή τι συνέπειες μπορεί να έχουν, αλλά όταν μιλάμε για τεχνικό έλεγχο είναι συγκεκριμένα τα πράγματα. Έτσι λοιπόν, με τη γνωμοδότηση αυτή, θα, αν και δεν μας λέτε αν πρόκειται για οδηγία ή κανονισμό. Ωστόσο, στο άρθρο 8, με μια τροπολογία σας, αναφέρεστε σε ορισμό. Εγώ ήξερα ότι ο ορισμός χρονικά πρέπει να μπαίνει στο διατακτικό, αλλά ε, εσείς τον ορισμό του βάζετε στο παράρτημα. Είναι αυτό σωστό, γιατί η περιοδικότητα του τεχνικού ελέγχου δεν υπάρχει στο κείμενο. Δεν θα πρέπει να το καλύψουμε αυτό. Επίσης, τα δεδομένα των κατασκευαστών το αναφέρετε κι εσείς, πρέπει να είναι διαθέσιμα για τον υπεύθυνο που προβαίνει στον τεχνικό έλεγχο. Αλλά θα λαμβάνονται υπόψη αυτή η τροπολογία υπαριθμών 9 οι ε, αντιπρόσωποι, των, οι ανεξάρτητοι αντιπρόσωποι, γιατί αναφέρεστε σε διάφορες κατηγορίες, αλλά όχι στον ανεξάρτητο αντιπρόσωπο. Και τρίτη και τελευταία ερώτηση. Όλα αυτά σχετίζονται με την εσωτερική αγορά. Δεν χρειάζεται μεταφορές να αναφερθούν ρητά. Μιλήσατε για αμοιβαία αναγνώριση και δοκιμές. Αλλά ο τομέας των μεταφορών έχει δικά του χαρακτηριστικά. Υπάρχουν χώρες ε, με μεγάλο τομέα μεταφορών. μπορούμε να τις θέσουμε στο ίδιο επίπεδο, σε ισότιμη βάση, με εκείνες των οποίο ο τομέας των μεταφορών είναι περιορισμένος. Ή μετά διαχωρισμοί όπως αν πρόκειται για ε, όχημα ε, ή για φορτηγό ή για δίκυκλο Όλα αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να τα συζητήσουμε πριν προχωρήσουμε περισσότερο. Ευχαριστώ κύριε Σμίντ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Από ό,τι φαίνεται είμαι παγίος αυτός που αντικαθιστά τους Τέλος πάντων, ίσως θα πρέπει αυτό να το βάλω στην κάρτα. Τέλος πάντων, ο κύριος ε, Μάντερ, τον οποίο στο σήμερα τις απόψεις και θεωρεί ότι η πρότασή σας είναι πάρα πολύ εύστοχη. Θα τις ψηφίσει. Θεωρεί ότι ευθυγραμμίζεται η έκθεσή σας με τη δική του. Επίσης ο κύριος Μάντες θέλει πολύ την αμοιβή αναγνώριση. Οπότε, νομίζω ότι θα υπάρχει ευρεία υποστήριξη των τροπολογιών σας, αλλά αυτό που θα ήθελα να πω τώρα αυτές είναι οι δικές μου απόψεις, είναι το εξή. Ξέρετε, στη χώρα μου, μόνο βουλευτής πολλά χρόνια, και εκεί θεώρησαν ότι πρόκειται για δοκιμή της επικουρικότητας. Τόσες φορές, 29 φορές το, το, το διεκδικήσαμε αυτό, κάναμε αυτή την ένσταση της υπηρετικότητας, είμαστε οι πρωταθλητές. Τέλος πάντων, αυτά είναι εσωτερικά μας θέματα. Δεν ξέρω όμως, μήπως αυτό το θέμα δεν σχετίζεται με δραστηριότητες διασυνοριακές, γιατί μου προξενεί κάπως έκπληξη το ότι έχουμε βεβαίως και <clears throat> διαφορετικές δυνατότητες και πρότυπα δοκιμής, τουλάχιστον έτσι πιστεύουμε, αλλά, αλλά αυτό το, όλο θέμα της κινητικότητας. Εντάξει, είναι θέμα ε, είναι θέμα αναγνώρισης όλων. Αυτό θα να είναι θέμα των αρχών της κάθε χώρας. Μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας. Καμιά φορά νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι έτσι αναπτύσσεται ακόμη περισσότερη κινητικότητα στην Ευρώπη. Και με αυτούς τους νόμους που φτιάχνουμε τελικά ε, στηριζόμαστε στις εθνικές αρχές και έτσι δημιουργούμε ένα κοινό ευρωπαϊκό πνεύμα. Ε, ο σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, ξέρω. Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσω ο κ. αλλά τα κάτι μέλη πάντω νομίζω θα προτιμούσαν οδηγία αντί κανονισμού. Λυπάμαι για τους ανθρώπους που τώρα ήρθαν, ότι αφιέρωσαν τόσο χρόνο στο πρώτο ζήτημα και οι συνάδελφοι που αργήσαν έχασαν την τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση. Τέλος πάντων, θα δώσω τώρα τον λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ιδιαίτερος εσάς προσωπικά για την έκθεση αλλά και τα μέλη της Επιτροπής σας. Πολύ χρόνο έχετε αφιερώσει, το ξέρω, στα θέματα αυτά. Έχετε μελετήσει τις συνέπειες, έχετε κάνει μια δεξιωτική συζήτηση. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο αφορά φυσικά την ε, ασφάλεια, την οδική ασφάλεια, αλλά και την εσωτερική αγορά. Νομίζω ότι πρέπει να δούμε τις πτυχές που σχετίζονται με την εσωτερική αγορά, πρόσβαση στα δεδομένα, πρόσβαση στην πληροφορία, η δυνατότητα για ε, προσφυγή σε ένα ανεξάρτητο συνεργείο και ηλεκτρονική μορφή του πιστοποιητικού. Πρόκειται για ζητήματα στα οποία Φαντάζομαι δεν έχετε ε, διαφωνίες με τον κύριο Κάρινς της ε, Επιτροπής Βιομηχανίας. Σαφήνεια λοιπόν και συνέπεια ως προς τη λειτουργία του κανονισμού, που είναι επίσης πολύ σημαντικά μέτρα. Η προσοχή του καταναλωτή, η αντιμετώπιση των ε, απατών σε σχέση με τα χιλιόμετρα, με τις τροπολογίες 12 και 14 για τις αναπροσαρμογές, τις παραποίησεις. Είναι πολύ ευπρόσδεκτες προτάσεις. Όλα αυτά ε, νομίζω ότι λίγο πολύ με αυτά που μας είχαν και εμάς ε, αποσχολήσει. Αλλά ένα σημείο που θα ήθελα να υπογραμμίσω που έχουν μια διαφοροποίηση είναι οι τροπολογίες 4 με 7. Εσείς μπορείτε να προτιμάτε την απλούστευση, ναι, αλλά για λόγους ε, λογικής θα πρέπει να διατηρήσουμε κάποιες ε, βασικές διατυπώσεις ώστε να ξέρουμε, να εξασφαλίσουμε ότι θα διαφυλάσσεται η ακαιρεότητα του αυτοκινήτου, του οχήματος. Δεν θα υπάρχει δηλαδή επέμβαση στην ακαιρεότητα του οχήματος. Να ξέρουμε ότι έχουμε να κάνουμε με το αρχικό, το αυθεντικό Διαφορετικά μπορούμε να καταλήξουμε να καλύπτουμε οχήματα που δεν έχουν καμία σχέση με το αυθεντικό. Επίσης τα δίτροχα με κινητήρα. Έχει αποφασιστική σημασία αλλά και η Επιτροπή Μεταφορών βεβαίω ενδιαφέρεται. Αλλά παρακαλώ τουλάχιστον δεχθείτε ότι μπορούμε να διαφωνούμε προς το παρόν. Αφήστε μας το περιθώριο να διαφωνήσουμε. Πάντως πρέπει να συμπεριληφθούν αυτή τη στιγμή, αυτή την εποχή τα δίτροχα με κινητήρα στο νομοθέτημα. Εάν τυχόν προκύψουν σοβαρά προβλήματα ως προς τον τύπο των δοκιμών που προβλέπονται και νομίζω ότι από τη συζήτηση έχουμε δώσει πολλές εξηγήσει ότι θα είναι ε, μόνο οπτική επαλήθευση, περιορισμένος ο έλεγχος και αν θέλετε και κάποια όριος προς τον κυβισμό λόγω της ε, χρήσης και τη συμπεριφορά του οδηγού, γιατί ανάλογα με το μέγεθος του κινητήρα είναι διαφορετική και η χρήση του, της μηχανής, ε, της μοτοσυκλέτας. Ε, αφήστε μας λοιπόν να το βάλουμε έτσι και αν έχετε αφιβολίες μπορούμε να τα ξαναδούμε. Τα στοιχεία μέχρι τώρα μας λένε ότι τα δίτροχα με κινητήρα έχουν πολύ παρόμοια συμπεριφορά κυρίως προς το περιεχόμενο της τεχνολογίας με τα τετράτροχα, με τα αυτοκίνητα δηλαδή, και θέλουμε να μπορούμε να κάνουμε τις σχετικές δοκιμές. Για τα σχόλια του κύριου Σμιτ, που είναι κάπως πιο προσωπικά, και θέλω και εγώ εδώ να δηλώσω ότι μιλάμε για μια πρόταση που αφορά ελάχιστους κανόνες. Βεβαίως πρέπει, ομολογούμε, να δοθεί ένα περιθώριο στην ευελιξία τα κράτη-μέλη. Αλλά έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο που χρειάζονται οι κανόνες. Και νομίζω ότι έχουμε βρει μια καλή ισορροπία. ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι αυτά τα που είπατε μπορούμε να τα λάβουμε υπόψη. Για τις τροπολογίες μέχρι 25 Μαρτίου έχουμε πρόθεσμη. Θα σκεφτώ αυτό που είπατε για τα ιστορικά οχήματα και να δούμε μήπως μπορώ να βάλω ε, μια επιπλέον διάταξη αλλιώς θα αφήσω τα πράγματα όσοι έχουν και όποιος θέλει μπορεί να αποβάλει τροπολογία. 24 ε, θα ζητεί και 25, 25 Απριλίου θα ψηφίσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστούμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και πάλι ρητώ συγγνώμη γιατί τόση ώρα συζητήσαμε το πρώτο θέμα και είμαστε, έχουμε, έχουμε χάσει μισή ώρα από το πρόγραμμά μας. Πέστε μου ποιος θέλει να φύγει για να προσπαθήσουμε να επιταχύνουμε. Γιατί δεν έχουμε ώρα. Βελτίωση τη πρόσβαση δικαιοσύνη Ευρωπαϊκή Ομοφωνία σε διασυνορικέ πολιτικέ εμπορικέ διαφορέ. Κύριε Ρόσφορντ είναι εδώ. Κύριε Πέρα, όχι. Ούτε ο κύριο Φόξ είναι εδώ. Για να δούμε τι έχει να μας πει. Ο κύριος Χάνς Πέτερ Μάγκερ έχουμε και εκπρόσωπο της Επιτροπής. Μάλιστα, μάλιστα. Γεια σας, καλώς ορίσατε. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή. Κατόπιν κύριο Ροσφόρ και κατόπιν ποιο άλλος θέλει. Και κατόπιν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Μάγερ, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, Μια έκθεση λοιπόν ευχάριστη. Αν συγκριθεί με το, την υπόθεση του, ε, της διαμεσολάβησης εμπορικές συναλλαγές, γιατί είμαι μόνος μου ε, ως εισηγητής και γενικά οι τροπολογίες που κατεθεί μου φαίνονται και ε, σύμφωνες με το ε, πνεύμα της δικής μου γνωμοδοτήσεις. Έχουμε από την κυρία Χοσφόχ 5, από την κυρία Ράπτη μία και από την Ισπανή συνάδελφο 8 τροπολογίες, 21 στο σύνολο είναι, και οι δικές μου βέβαια, είναι συμπλήρωμα και ε, βελτίωση της ε, γνωμοδότησης, της υποστηρίζω και της 21 ιδιαίτερα δε εκείνες που ζητούν ε, μια καλύτερη εκστρατεία ενημέρωσης με, κατανο... με κατανοητά στοιχεία και πληροφορίες και κυρίως περαιτέρω μέτρα κατάρτισης των επαγγελματιών, δικηγόρων κτλ. Αν και εδώ θα έλεγα ότι καλό είναι να μην αναφέρουμε συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών. Το ευεργέτημα της παινίας έχει συγκεκριμένες οριακές τιμές, οι οποίες εξίσου ισχύουν για τον κάθε ενδιαφερόμενο ανάλογα με το εισόδημά του είτε έχει επαγγελματική δραστηριότητα μια κατηγορία, είτε, κατηγορίας, είτε όχι. Δεν πρέπει δηλαδή να κάνουμε διαφοροποίηση προς, το θέμα αυτό, γιατί ισχύει ο ίδιος, ε, ε, η ίδια νομοθεσία για κάθε πολίτη. Όσον αφορά το ευεργέτημα της ε, παινίας στις ποινικές διαδικασίες δεν θεωρώ ότι έχουμε αρμοδιότητα, είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών, είναι το ποινικό δίκαιο ακόμη και στη διασυνοριακή του διάσταση και ως εκ τούτου πιστεύω ότι πρέπει να το αγγίξουμε. Από την άποψη του ποινικού δικαίου το μόνο που θα μπορούσαμε να κάνουμε θα ήταν αν υπάρχουν ζητήματα συγκεκριμένα προβλήματα όπως σε παραδείγματι αυτό των, ε, της των δικαιωμάτων του δημιουργού κτλ. Να ζητήσουμε την ποινικοποίηση από πλευράς των κρατών μελών της ε, παραβίασής τους. Όχι ακόμα όμως. Η κυρία Ράπτη έχει κάνει μια τροπολογία εδώ. Ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με, το, με τη μετάβαση τα έξοδα σε μια πρώτη προσέγγιση στον δικηγόρο, θα έλεγα το προκαταρκτικό στάδιο, πριν φτάσει κανείς στο δικαστήριο δηλαδή. Συνήθως ακόμη και σε διανοσυναριακές ε, συναλλαγές μπορεί κανείς να βρει δικηγόρο και ε, στην χώρα του με ελάχιστο κόστος ε, μετάβασης, αλλά Εάν χρειαστεί κανείς να ταξιδέψει για να παραστεί σε μια κροματική διαδικασία, εάν έχει προσκληθεί με προσωπική κλίση και πρέπει να ταξιδέψει σε άλλο κράτος, αλλά τότε μόνο μπορούμε να συζητήσουμε, αλλά εάν ε, τότε μόνο συζητούμε την ε, δυνατότητα αποζημίωσης των εξόδων, τότε βρισκόμαστε σε ένα πεδίο άνισο, γιατί θα σήμαινε αυτό ότι πριν από την έγκριση των εξόδων με βάση το ευεργέτημα της ποινίας προεξοφλούμε την έκβαση μιας δίκης. Και έτσι θα έλεγα ότι το πιο σωστό είναι εφόσον προσφέρονται έξοδα δίκης με το ευεργέτημα της ποινίας, σε αυτά θα καλύπτουμε και την μετάβαση, την ε, κίνηση. Επίσης θα πρέπει να στήσουμε από τα κράτη-μέλη να βελτιώσουν τις διατυπώσεις, να ενημερώσουν με μια ευρύτατη διαδικασία εκστρατεία ενημέρωσης. Πολλοί από εμά που έχουμε εργαστεί στο νομικό, στο κλάδο του δικαίου, ξέρουμε πόσο αξιοθρύνητη είναι η κατάσταση σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά το ευεργέτημα της παινίας. Σας ευχαριστώ πολύ. κυρία Βάιλερ, αντί για την κυρία Ράπτη όχι. Ο κύριος Ροσφόρ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Και όπως και ο κύριος Μάιερ, θα ήθελα να επισημάνω ότι έχουμε μια εξαίρετη γνωμοδότηση με εξαίρετο συντάκτη. Μόλις, τη λέξη, μόλις είπα τη λέξη ραπορτέρ, βάλατε και τα ακουστικά σας. Εξαιρετικός ο συντάκτης. Και αυτό το λέω για να δείξω το συνενετικό πνεύμα το οποίο ξεκινάει η συζήτηση και συμφωνώ με το όσο είπε ο κύριος Μάγερ για την ενσωμάτωση μιας ποινική διάστασης στην υπόθεση αυτή, που τους άλλους δεν θα ήταν και αρμοδιότητα της δικής μας Επιτροπής. Ταυτόχρονα, όπως είπε και ο κύριος Μάγερ, ότι με πολύ συμπάθεια βλέπει τις ε, τροπολογίες των συναδέλφων, γιατί και εγώ βλέπω ότι οι δικές του τροπολογίες βελτιώνουν το κείμενο, τις υποστηρίζω συνολικά ο κύριος Μάγερ σωστά καθιστά πιο σαφές και ακριβές το κείμενο ως προς την θέσπιση μιας ευρωπαϊκής ομάδας δικηγόρων που θα μπορούσε να αντιδράσει. Και μας λέει ότι σε αυτή την ομάδα θα μπορούσαμε να βρίσκουμε δικηγόρους που μιλούν τη γλώσσα και έχουν την εξειδίκευση για το δικαιικό σύστημα που ζητείται. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί η αξιολόγηση που έχει γίνει της εφαρμογής οδηγίας δείχνει ότι υπάρχουν πρακτικές δυσκολίες ως προς την ε, σωστή ε, εφαρμογή του δικαίου. Και έτσι νομίζω, όπως συμβαίνει και στη χώρα μου, ότι μπορούμε να ορίσουμε μία μόνη αρχή, κράτος μέλος, μία μόνη μονάδα συγκεκριμένα που θα δέχεται τα αιτήματα για ε, το πλεονέκτημα της παινίας, μία μονάδα για κάθε κράτος μέλος. Ενιαία πάντως. Και ο κύριος Μάγερ πολύ σωστά είπε τώρα ότι για να ενισχυθεί η ενημέρωση και το άρθρο 18 βεβαίως της οδηγίας πρέπει να γίνουν όλα αυτά. Εγώ στην ανταλλαγή απόψεων στις 21 ε, Φεβρουαρίου είχα ε, προτείνει κάποιες τροπολογίες. Θα επισημάνω μία-δύο για την ε, διάσταση των προτάσεων Διερωτώ με. Στο ε, ερωτηματολόγιο, αν το θεωρεί πιο ευανάγνωστο με το τύπο Word που αναφέρει ο εισηγητές, μα είναι σωστό όμως εμείς να λέμε να ονομάζουμε ένα συγκεκριμένο λογισμικό και μάλιστα αυτό που γνωρίζουμε ότι ανήκει σε μια ε, αμερικανική εταιρεία που έχει και μονοπωλιακή στάση και συμπεριφορά στην υπόθεση αυτή, ενώ υπάρχουν και άλλου τύπου, άλλα αντίστοιχα λογισμικά που μπορούν να αξιοποιηθούν. Δεν θα ήταν πιο απλό να αποσυρθεί ή μη τι άλλο η συγκεκριμένη αναφορά σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα λογισμικού, πρόγραμμα που ανήκει σε μια εταιρεία. Επιμένω και στο θέμα των ε, οικονομικών κριτηρίων. Θα επανέλθω όπως τα έχω αναφέρει ήδη. Όχι λόγω υπερβάλλοντος ζήλου, αλλά γιατί ε, το κόστος ζωής στην κάθε χώρα είναι διαφορετικό. Υπάρχουν ερμηνείες διαφορετικές ανάλογα με το κράτος ε, προέλευσης και το κράτος της ε, αρμόδιας αρχής, η οποία θα μπορούσε να απαγορεύσει ή να μην λάβει υπόψη τα οικονομικά κριτήρια. Όπως και να έχει, εγώ δεν θα ήθελα να αφήσουμε τα πράγματα στην τύχη, να είμαστε δηλαδή πιο συγκεκριμένη, ώστε ό,τι είναι να λαμβάνετε υπόψη στο δυνατόν πιο σωστά. Και θα ήθελα να αναφέρω και κάτι σχετικό με την ε, ε, τροπολογία της κυρίας Ράπτη που ανέφερε και ο κύριος ε, Μάγερ. Πρέπει να πω ότι όταν τη διάβασα την τροπολογία αυτή, ξαφνιάστηκα δεν ήξερα πώς να την ερμηνεύσω, γιατί ίσως να μπορεί να εννοεί αυτή η τροπολογία ότι πρέπει να καλύπτουν τα έξοδα μιας πρώτης επίσκεψης μετάβασης πριν από την εφαρμογή, την απόφαση για εφαρμογή του ευαργήματος της παινίας και χωρίς να ξέρουμε τι μοίρα θα έχει αυτό το αίτημα εάν υποβληθεί. Δηλαδή είναι σαν να γνωρίζουμε ευεργέτημα της παινίας προκαταβολικά ή αλλιώς γίνεται αναδρομικά αυτή η ε, αποζημίωση. Δίνεται αναδρομικά αυτή η αποζημίωση. Εκεί μπορώ να το δεχθώ. Αλλά να προεξοφλούμε ότι θα χορηγηθεί το, το ευεργέτημα της παινίας μου φαίνεται πολύ δύσκολο. Αυτό ήταν που με απασχολούσε προς την τροπολογία της κυρίας Ράπτη. Δεν είμαι πεπισμένος όπως έχει τώρα η κατάσταση. Α ας μας πει ο κύριος Μάγερ. Γιατί περιμένω και περιμένω να ακούσω βέβαια και την άποψη της Επιτροπής με αδημονία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πιστεύω ότι μπορούμε να τελειώσουμε τη δουλειά αυτή αποτελεσματικά μεταξύ μας. Μην ξεχνάμε ότι ο στόχος μας είναι, με τη γνωμοδότηση αυτή, να δώσουμε ενάψματα για σκέψη στην αρμόδια κατουσία επιτροπή, που είναι η Επιτροπή των Νομικών Υποθέσεων. Ευχαριστώ. Θέλει κανείς άλλο το λόγο. Αν δεν συγκρατήσετε άλλο, κύριε Ροσφόρ, ας ακούσουμε την Επιτροπή πολύ γρήγορα να μας πει τι γνώμη έχει. Ε, thank you very much. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε είμαι σύντομη. Να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας για το ενδιαφέρον σας όσον αφορά την οδηγία για το ευεργετήμα παινίας. Ναι, είναι κάτι το, που αφορά τους διαδίκους, για το αστικό δίκαιο, δεν αφορά τις ποινικέ δίκες. Μελετήσαμε την εκθεσή και συμφωνούμε για το πόσο σημαντικό είναι αυτή η επεκπαίδευση, τα μέτρα ενημέρωσης για ε, τις σχετικές τροπολογίες, τις λάβουμε υπόψη. Επίσης όσον αφορά τη βελτίωση για την ενημέρωση όσον αφορά τις ε, διαδικτυακές υπηρεσίες στις δικαιοσύνη. Για το, το δίκτυο αυτό, αυτό τον ιστότοπο, αυτά που προβλέπονται στο άρθρο 18 της οδηγίας, το οποίο αναφέρει και η έκθεση. Βεβαίως και θα ληφθεί και αυτό υπόψη. Τώρα, δεν θέλω να επισέλθω σε λεπτομέρειε ακόμη, Απλώς να σας ευχαριστήσω για τις απόψεις σας. Και όταν δώσουμε συνέχεια στην ε, έκθεση θα σας ε, λάβουμε υπόψη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μάγερ. Θέλετε κάτι να προσθέσετε. Μάγερ. Πολύ σύντομα. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλά δυσκολίε στη Γερμανία για, το, για την ομάδα των δικηγορών. Υπάρχει ήδη η δυνατότητα της επικοινωνίας μέσα του διαδικτύου και από εκεί ήδη μπορεί να διευκρινιστεί ή να εξευρεθεί ένας δικηγόρος ο οποίος έχει γλωσσικές γνώσεις, γαλλικά, ισπανικά κτλ σωστό είναι αυτό που λέτε για την αναφορά σε μια εταιρεία ή σε ένα λογισμικό συγκεκριμένη εταιρεία. Απλώ εννοούσα ότι θέλω ένα απλό λογισμικό που μπορεί κανεί να συμπληρώσει, γιατί πολύ συχνά όταν ε, πρέπει κανεί να συμπληρώσει ένα έντυπο ε, στο για το ευεργέτημα της παινίας κάνοντας το ενέτησή του ε, να μην βρίσκει τον τρόπο, δηλαδή χρειάζεται να κάνει πληρωματικές ερωτήσεις, να απαντήσεις πληρωματικές ερωτήσεις κτλ. Αυτό που εννοώ λοιπόν εγώ είναι να μπορεί να, ότι πρέπει να μπορεί να κατεβάζει κανείς το έντυπο, να μπορεί να το αποθηκεύει, να είναι εύχριστο. Και ως εκ τούτου παρακαλώ και την Επιτροπή όταν επαληθεύει τα έγγραφα, αυτά τα έντυπα δηλαδή, να ακολουθεί ε, την ίδια απεικόνηση για το έντυπο ανεξαρτήτως γλώσσας. Όχι απλώς δηλαδή το ίδιο περιεχόμενο, αλλά την ίδια απεικόνηση, να μην υπάρχει διαφορά στην ε, οθόνη ανάλογα με το ποια γλώσσα χρησιμοποιώ. Γιατί έτσι είναι πολύ πιο εύκολο, ε, ακόμα και αν ε, βρίσκομαι σε μια γλώσσα την οποία δεν κατέχω πολύ καλά, να ακολουθήσω τη σειρά και να συμπληρώσω. Νομίζω ότι αυτό έχει μεγάλη σημασία για τον καταναλωτή. Χαίρομαι που μπορούμε να ε, διαπιστώσουμε εδώ γενικά ε, συμφωνία, συνένεση. Σας ευχαριστώ. Έχουμε τις τροπολογίες σας, τις οποίες θα ψηφίσουμε την 10η Απριλίου. Θα ψηφίσουμε την πρόταση στη διάρκεια του Μαΐου, επομένως. Ευχαριστούμε πολύ. Προχωράμε λοιπόν στο τελευταίο μας θέμα για τη σημερινή μας συζήτηση. Έχουμε εδώ και εκπρόσωπα της Επιτροπής και θα συζητήσουμε την ισόρροπη εκπροσώπηση των φίλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητών στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών. Χαίρομαι διότι βλέπω ότι η κυρία Αντωνία Παρβανόβα είναι εδώ. Δεν η κυρία Χερδέν είναι εδώ. Για να δω λίγο ποιοι άλλοι έχουν μείνει. Η κυρία Βάιλερ. Θα μιλήσετε εξ ονόματος της κυρίας Χαίδησης, κυρία Βάιλερ. Ο κύριος Μπίλερ είναι εδώ. Νομίζω ότι έχουμε ε, όλες τις ομάδες και εγώ θα κάνω... Ε, όχι, έτσι λοιπόν αφού ο κύριος Μπίλερ είναι εδώ θα κάνω εγώ σχόλια. Λοιπόν, ε, υπάρχει κάποιος από την Κομισιόν. Πολύ ωραία. Μήπως θα μπορούσατε να μας πείτε ποια είστε, γιατί δεν σας βλέπω στον κατάλογό μου. Είμαι η ε, υποδιευθύντρια του τμήματος ε, ισότητας ε, της ίσης μεταχείρισης ίσης μεταχείρισης στην Κομισιόν. Συγγνώμη που δεν ε, ε, ήμουν στον κατάλογό σας. Βάντερ Βλής λέγομαι. Βάντερ Βλής. Και Ρόσλιν το μικρό σας. Χαίρομαι πάρα πολύ Ρόσλιν. Η κυρία Παρβανόβα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η γνωμοδότηση αυτή αφορά μια πάρα πολύ θεραλέα ε, πρωτοβουλία της Επιτρόπου reading, που έχει ήδη κυκλοφορήσει μεταξύ των ε, εμπλεκομένων φορέων και των κρατών ε, μελών. Πολλές ήταν οι προηγούμενες πρωτοβουλίες οι οποίες αποσκοπούσαν στην βελτίωση της παρουσίας των γυναικών στα, σε, στα διοικητικά συμβούλια και τα εκτελεστικά συμβούλια. Ε, μέσα από μια διαδικασία αυτοελέγχου, η οποία όμως δεν έδωσε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ε, πιστεύουμε εμείς ότι περισσότερες γυναίκες σε θέσεις διοικητικών στελεχών μπορούν να βελτιώσουν την αποδοτικότητα της επιχείρησης. Ε, αλλά χρειάζεται η λήψη συγκεκριμένων μέτρων, μια και τα εθελοντικά μέτρα δεν κατάφεραν να μειώσουν, να κλείσουν αυτήν την ε, ποιοτική, αυτό το ποιοτικό χάσμα. Το θέμα των ποσοστώσεων είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Ε, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο της προηγούμενου μήνα υπάρχει μεγάλη ε, διαφορά. 49% ε, των ερωτηθέντων λένε ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η υποχρεωτική νομοθεσία. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και οι απλοί πολίτες μας πιστεύουν ότι μόνο με συγκεκριμένη εξαναγκαστική κατά κάποιο τρόπο νομοθεσία μπορεί κανείς κανείς να επιτύχει καλά αποτελέσματα. Ε, προσπάθησα να ε, παρουσιάσω ένα ισορροπημένο κείμενο το οποίο λαμβάνει υπόψη στοιχεία όπως είναι η νομική ασφάλεια για τις ε, επιχειρήσεις, η εσωτερική αγορά και οι ίδιες οι προτιμήσεις στη διάρκεια της πρόσληψης περισσότερες γυναίκες σε θέση διηγητικών στελεχών μπορούν ε, να βελτιώσουν περισσότερο, να επηρεάσουν περισσότερο τις επιλογές των αναγκών, γνωρίζουν ίσως καλύτερα δε, τις ανάγκες των καταναλωτών. Ένα άλλο ε, σημείο σημαντικό είναι η νομική ασφάλεια για τις κυρίως τις επιχειρήσεις αυτές οι οποίες ε, έχουν έδρα σε πολλές χώρες μέλη σε μερικές περιπτώσεις ε, η πολυπλοκότητα ή η διαφοροποίηση μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στην ε, σωστή λειτουργία των ε, επιχειρήσεων αυτών στις διάφορες χώρες και επομένως θα πρέπει να υπάρχει η απαραίτητη νομική ασφάλεια και οι κανόνες αυτοί οι οποίοι οικονομικά τελικά δεν θα αποβούν ζημιογόνες για την ίδια την επιχείρηση. και μελέτες της Deutsche Bank και άλλων ε, έχουν καταδείξει ότι ε, είναι προς το συμφέρον της εταιρείας από κάθε κατεύθυνση και από κάθε πλευρά και άποψη να έχει περισσότερες γυναίκες σε θέση διοικητικών στελεχών. Μας ενδιαφέρει η ισορροπή προσώπηση αλλά μια ε, καλύτερη παρουσία των γυναικών στα, στις θέσεις διοικητικών στελεχών μπορούν να βελτιώσουν ακόμα και την οικονομική ανάπτυξη της ε, εταιρείας. Σε περιόδους δημογραφικής κρίσης ε, ε, είναι σημαντικό να μην αφήνουμε ανεκμετάλλευτο το δυναμικό το οποίο ε, ε, προσφέρει το 50% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα ανθρώπινο κεφάλαιο το οποίο είναι στην διάθεσή μας το να έχουμε σωστούς υποψηφίους άντρες και γυναίκες για σημαντικές θέσεις θα βελτιώσει και την τελική επίδοση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. In και ε, βεβαίω μα ενδιαφέρει μέσα από τι θέσει των υψηλών διοικητικών στελεχών να έχουν ε, μεγαλύτερη πρόσβαση οι γυναίκε ε, και στις, στα δίκτυα τα οποία δημιουργούν οι γυναίκε, έτσι ώστε να είναι και πιο αποτελεσματική η παρουσία των, των γυναικών. Βεβαίω εδώ θα περιμένω και ένα input από του υπολείπου, αλλά εμεί πιστεύουμε ότι η απουσία γυναικών από τα θέσει εκτελεστικών στελεχών ε, είναι κάτι αρνητικό. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε τον πρόεδρο. Ποιος θέλει το λόγο. Η κυρία Λεγκρίπ. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Και εγώ με τη σειρά μου θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόταση αυτή της οδηγίας ε, του Νοεμβρίου. Θεωρώ ακριβώς όπως έχει δείξει και η συζήτηση είναι θέμα πάρα πολύ καυτό και έτσι θα γίνουν βήματα πρόοδου ουσιαστικά. Ανεξαρτήτως το τι μορφή θα λάβουν οι γελουρικές μας εργασίες για να διεκπαιρεώσουμε το θέμα. Είναι πολύ ενδιαφέρον το ζήτημα. Και ακριβώ είναι πολύ τολμηρό το κείμενο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι ουσιαστικό ζήτημα η συμμετοχή, εμπλοκή των γυναικών στα κέντρα αποφάσεων. Το θέμα είναι επίκαιρο, αφορά όλους τους τομείς του δημοσίου βίου. Οπότε να δούμε με ποιο τρόπο θα βελτιώσουμε την κατάσταση. Είναι λογικό επομένως το ότι και εμείς προσπαθούμε να δούμε τι θα γίνει όσον αφορά τα διοικητικά συμβούλια των μεγάλων εταιριών, όσον αφορά τη συμμετοχή των γυναικών. Κάνουμε διορθώση πορεία, να κάνουν προτάσει στα κράτη-μέλη, να αρθούν οι ανισότητες. Πολλές φορές είναι πάρα πολύ έντονες. Δεν χρειάζεται να υπάρχουν. Εξηγούνται βέβαια. Αλλά δεν υπάρχει λόγος να υπάρχουν τέτοιες ανισότητες. Άλλωστε έχουμε και όλες αυτές τις μελέτες που έχουν γίνει από πάρα πολύ σοβαρά γραφεία και καταδεικνύουν ότι όταν αρθούν αυτές οι ανισότητες λειτουργούν πιο εύρυθμα οι επιχειρήσεις. Και γι' αυτό και εμείς έχουμε ως στόχο να άρουμε αυτή την ανισότητα. Κυρία Παρβάνοβα, ασχολήθηκε με τα ζητήματα τα οποία είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής μας, της ΣΥΜΚΟ. Πώς δηλαδή θα βελτιωθεί η κατάσταση για τους ανθρώπινους πόρους στις επιχειρήσεις, πώς θα αρθούν όλες αυτές οι ανισότητες που αφορούν τελικά φραγμό όσον αφορά τη δραστηριότητα της επιχείρησης στην εσωτερική αγορά. Euh, και επομένως και εμείς θα δούμε πώς μπορούν τα πράγματα να κινηθούν με πνεύμα σύγκλησης, σε ένα πλαίσιο εναρμόνισης. και αντιστοίχω να διορθώσουμε και τις συνθέσεις στα διοικητικά συμφούλια. Το 2011 η Γαλλία εθέσπισε ένα νόμο προτάσει δύο βουλευτών ήταν πρόταση ιδίας νομοθετικής πρωτοβουλίας αυτών των βουλευτών η κυρία Μερμάν, και Σκοπέ, σκοπεύουν είναι από το δικό μου κόμμα, τη δική μου πολιτική οικογένεια προέρχονται και μετά από την προβληματική που αναπτύχθηκε έθεσε πίστη με αυτόν τον νόμο ένα σύστημα ποσοστώσεων που προβλέπουν 40% συμμετοχών στα διοικητικά συμβούλια των εταιριών που είναι συγκεκριμένε στο χρηματιστήριο. Και από τότε που ετέθησε ισχύ αυτός ο νόμος, αυτός του 2011, διαπιστώνεται μία αύξηση 15% της εκπροσώπησης των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια. Έχουμε δε καθορίσει ε, κάποιους ενδιάμεσους στόχους 2014 μέχρι το 2020 και ουσιαστικά ξεπεράσαμε το, το, το, πλάνο κάλυψης κάποιων ποσοστών. Τον Ιούνιο του 2012 έχουμε τα αντίστοιχα στοιχεία για το σύνολο των γαλλικών επιχειρήσεων όπου είχαμε εκπροσώπηση 23%. Και όσον αφορά τις 40 πιο μεγάλες επιχειρήσεις είχαμε 25,2% Συμμετοχή και εκπροσώπησης γυναικών στα διοικητικά συμβούλια. Σε εταιρείε του ΚΑΚ 40, 40 πιο μεγάλες. Και αυτό ήταν καθαρά αποτέλεσμα της αλλαγής της νομοθεσίας. Δεν λέω ότι θα πρέπει να κάτσουμε για να αντιγράψουμε ακριβώς τον ε, γαλλικό νόμο. Ναι, ναι, υπάρχουν πάντως έντονες διαφορές, ανισότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που απορρέουν από διαφορετικές ιστορίες, πρακτικές, ε, επαγγελματικέ, επιχειρηματικέ, παραδόσεις του κάθε κράτους οπότε και θα πρέπει να γίνεται κάθε φορά η διάκριση, η διαφοροποίηση και να βρεθεί μια ισορροπία μεταξύ της, του, τι θέλουμε να πετύχουμε και, και, τι, θέλουμε να επιβάλλουμε. Για άλλη μια φορά χαιρετίζω την επιμονή της ε, Επιτρόπου Ρέντινγκ. Ότι δηλαδή από τη μία μεριά ε, είναι δυναμική αυτή η ρύθμιση, αλλά από την άλλη μεριά αφήνεται το περιθώριο κριτική ευχαίρεια στα κράτη-μέλη για τον τρόπο με τον οποίο θα πετύχουν αυτό το στόχο ανάλογα με τα ιδιότυπα χαρακτηριστικά κάθε χώρας, κάθε κλάδου, κάθε περιοχής. Και η ισορροπία ακριβώς είναι η προσαρμογή του στόχου στις ιδιορυθμίες κάθε κράτους. υπάρχουν στόχοι επομένω με συγκεκριμένα ποσοστά, συγκεκριμένε ποσοστώσει. Αυτό θεωρώ ότι είναι αποτελεσματικό. Επομένω, αυτά τα οποία προβλέπουν θα πρέπει να τα υλοποιήσουμε στην Ένωση. Σε αυτή τη φάση δεν θα επισέλθουμε στις λεπτομέρειες γιατί θα το ξανασυζητήσουμε. συζητήσουμε για, για τα εκτελεστικά στελέχη των διοικητικών Συμβουλίων και τα μη εκτελεστικά. Ε, δηλαδή θα πρέπει να στείλουμε το πολιτικό μήνυμα που θέλουμε για την ισότητα. Από την άλλη μεριά βέβαια θέλουμε το μια προς επιχείρηση είναι ότι δεν θέλουμε να, να θεσμοθετηθεί μια παρέμβαση ε, όσον αφορά την διαχείριση των εταιρικών θεμάτων. Τέτοια ισορροπία θα πρέπει να βρούμε. Και το κείμενο θα εμπλουτιστεί, θα τροπολογηθεί κατόπιν των κοινοβουλευτικών εργασιών. Ένα κείμενο ισορροπημένο επομένω. Το οποίο θα μας βοηθήσει να πετύχουμε το στόχο μας. Θα πρέπει να τον πετύχουμε. Καλύτερη περισσότερη παρουσία, περισσότερη εμπλοκή των ε, γυναικών σε όλους τους τομείς του δημοσίου, του οικονομικού βίου. Αυτό είναι το διακύβευμα ε, γιατί θα, έχουμε περισσότερη ανταγωνιστικότητα και θα είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Ευχαριστώ. Πολύ χρήσιμη η συμβολή σας. Να δούμε τι θα συμβεί στη Γαλλία. Θα παρακαλέσω την κυρία Βάιλερ να μας πει τη γνώμη της τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι όντως πολύ ενδιαφέρον να βλέπουμε όλες τις χώρες, όχι και την Νορβηγία βεβαίως, και το όσα συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια, αλλά και όσα δεν λαμβάνουν χώρα. Συμφωνώ με τους και τις προλαλήσαντες και προσλήσαντες. Δεν πρέπει, κυρία Λεγκρή, να είμαστε πολύ ψοφοδείς. Βεβαίως να σεβόμαστε και να ακούμε και τα λοιπά, αλλά με ποσοστώσεις και δεσμεύσεις δεν προχωράμε πολύ. Νορβηγία, Γαλλία, Σκανδιναβία, όλοι οι εμπειρία όλων των κρατών δείχνουν ότι χωρίς ε, δεσμευτικούς όρους δεν κάνουμε τίποτα ως προς τις ε, ποσοστώσεις. Γι' αυτό συμφωνώ με την ανάλυση βλέπω κάποιες παρατηρήσεις τις οποίες θέλω να υποβάλω στον εισηγητή, σας τις διαβάζω γιατί μου φαίνεται και εμένα πολύ ενδιαφέρον. Κάποιοι λένε ότι κάποια κράτη-μέλη, συμπεριλαμβανομένου και του οικείου, δεν έχουν συστήματα δημόσιας ανακοίνωσης ελεύθερων θέσεων και θα ήθελε διαδικασία διαφανή και ουδέτερη. Διαφορετικά δεν μπορεί κανείς να έχει ε, την ευκαιρία για την ενημέρωση και την πρόσβαση. Επίσης χρειάζεται μία ε, δυνατότητα για υποβολή προσφυγών σε περίπτωση που κάτι δεν έχει λειτουργήσει σωστά Θέλει να υπογραμμίσει επίσης το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Είναι σημαντικό να υπαχθούν και οι μεγάλες μη εισηγμένες εταιρείες να μπουν στο πεδίο εφαρμογή, γιατί ξέρουμε ότι η κυρία Βόητοβα είχε πει να μην, ε, είναι η μεγάλη, να μην επαγόνται οι μεγάλε επιχειρήσει. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει και οι μεγάλε επιχειρήσει. Στο τελευταίο σημείο αναφέρατε στις διακρίσεις. Εσείς, κυρία Παρβάνοβα, αναφερθήκατε σε κυρώσεις με τη μορφή χρηματικής ποινής. Δυνατόν, πιθανόν και αυτό. Αλλά ίσως και άλλες κυρώσεις να είναι δυνατές είναι απαραίτητο να υπάρξουν αυτές οι προτάσεις. Ε, αυτά ήθελα να πει στην, ε, συντάκτρια. Κλείνοντας, ήθελα να πω ότι θα ήμουν πολύ ευτυχή αν μπορούσαν να δώσουν οι γυναίκε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα σαφέ μήνυμα πριν από την προσεχή εκλογική αναμέτρηση και πιστεύω μπορούμε να τα καταφέρουμε. ότι έχουν σημασία. Έχει σημασία να εξασφαλιστούν οι ώρες της ε, συμμετοχής και των εφιών γυναικών, όπως και των εφιών ανδρών, γιατί δεν θέλουμε να τους αποκλείσουμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για αυτές τις ενθαρρύνσεις. Να πω και εγώ δύο λόγια σαν σκιώδης από την ομάδα μου. Πρώτα απ' όλα, δεν χρειάζεται να με πείσει κανείς για το ότι θα πρέπει περισσότερες γυναίκες να συμμετέχουν ε, σε θέσεις διηγητικών στελεχών. Είναι γεγονός ότι δεν ε, εκμεταλλευόμαστε ε, το δυναμικό ενός τμήματος του πληθυσμού που έχει γνώσεις και είναι καλά εκπαιδευμένο. Νομίζω ότι άλλωστε πρέπει να αλλάξει όλη η πρακτική πρόσληψης ε, υπαλλήλων και πρόθεση καριέρας. Όλα αυτά λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικά. Με, ποια, με μια έννοια, συμφωνώ με την κυρία Χέντου, ότι θα πρέπει να βάλουμε, ε, να κάνουμε συγκεκριμένες ε, τροποποιήσεις, αλλά πρέπει να σας πω ότι δεν πείθομαι καθόλου ότι στρατηγικές απαιτήσει μπορούν να ε, αφορούν μονάχα τις συσυγμένε στο χρηματιστήριο. Βεβαίως θα μπορούσε να είναι ένα μήνυμα, αλλά δεν είμαι σίγουρη για την αποτελεσματικότητα. Πιστεύω ότι θα είναι δύσκολο να επιβληθεί κάτι τέτοιο. Οι κυρώσεις που ζητούνται, τι είναι, διοικητικά πρόστιμα, να, ίσως αλλά και αναφέρεται ότι ενδεχομένως μπορούν να υπάρξουν και άλλα συνοδευτικά μέτρα κτλ. Δεν νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπίσει κανείς το θέμα αυτό. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι πολλά μπορούν και πρέπει να γίνουν από την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χαίρομαι που η κυρία Ρέντιγκ ανέλαβε αυτή την ε, πρωτοβουλία και όπως είπε η κυρία Παρβάνοβα ε, μεγάλο αντίκτυπο είχε η πρωτοβουλία αυτή. Θα πρέπει να δοθούν πάντως περισσότερα στοιχεία. Θα γίνουν περισσότερες μελέτες περιπτώσεων έτσι ώστε να ε, δοθούν πρότυπα και role models για γυναίκες, νέες γυναίκες, οι οποίες μπαίνουν τώρα στην αγορά εργασίας ή μπαίνουν για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας, έτσι ώστε να αλλάξουν στάσεις, απόψεις, νοοτροπίες. Ε, η εστίαση σε μια συγκεκριμένη κατηγορία εταιριών δεν νομίζω ότι βοηθάει στην πρόθεση του ζητήματος. Αυτή είναι η δικιά μου οπτική γωνία. Εγώ νομίζω ότι θα είχα μια άλλη προσέγγιση. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν και κάποιες απόψεις ε, οι οποίες εύκολα μπορούν να ε, απορριφθούν Ας πούμε, στον Ηνωμένο Βασίλειο, νέες προσλήψεις σε μεγάλες εταιρείες δείχνουν ότι 36% στις μεγάλες, γυναίες, στις μεγάλες εταιρείες ε, ε, καλύπτονται από γυναίκες και αυτό το ποσοστό πέφτει στο 32% στις μικρότερες εταιρείες. Αυτό νομίζω ότι είναι ενθαρρυντικό. Τώρα το να βάλει κανείς σε ποσόστο 40% για όλες τις επιχειρήσεις και τις εταιρείε. δεν ξέρω αν είναι ο καλύτερος τρόπος. Η κατάσταση έτσι όπως διαμορφώνεται είναι ενθαρρυντική και μας δίνει κάποια θετικά μηνύματα. Αυτή είναι η θέση της ομάδας και νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε και κάποια άλλα ε, θέματα, έτσι ώστε να μπορέσουμε και από άλλες πλευρές να βελτιώσουμε τη θέση των γυναικών. Κάποιος άλλος θέλει να μιλήσει. Όχι. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Βάντερ Φλής ε, να μας πει δύο λόγια. Καλώς ορίσατε. Είναι η πρώτη φορά που είστε στην Επιτροπή μας. Σας ευχαριστώ πολύ για το θερμό καλωσόρισμα. Είναι μεγάλη μας χαρά Επιστώνουμε ότι ενδιαφέρεται εντόνως η Επιτροπή σας για αυτή τη σημαντική πρόταση και ιδιαιτέρως θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την εισηγήτρια, την κυρία Παρβάνοβα για τον ενθουσιασμό με τον οποίο αγκάλιασε το θέμα, για τα, όσα ανέλησε για το, για το ζήτημα, το οποίο βεβαίω και είναι μια πάρα πολύ καλή αρχή. Ε, και εμείς αντιστοίχως αποφασίσαμε να κατεβάσουμε την πρόταση ε, προς εσάς να το εισηγηθούμε ε, και προς το Συμβούλιο. Τώρα θα ήθελα να σας αναφέρω ε, το ιστορικό πλαίσιο αυτής της ε, πρότασης και κατόπιν να θίξουμε τα ζητήματα τα οποία είπα, ανέφεραν και οι αγορητές και επανειλημμένα ανεφέρθη ότι ε, και εσείς το είπατε κυρία Λεγκρίπ ότι οι ποσοστώσεις κάθε αυτέ δεν σα ενδιαφέρουν, αλλά τα αποτελέσματα είναι αποτελεσματικά. Δηλαδή, αυτό είναι το ζήτημα, ότι η ισότητα των ε, φύλων είναι μία από τι ε, βασικές αξίες θεμέλιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επομένω για αυτό το ζήτημα έχουμε προσπαθήσει με διάφορε πρωτοβουλίε να νομοθετήσουν. Καμιά φορά είχαμε και την αυτορύθμιση, η οποία δεν επέτυχε. Είχαμε κάποιε συστάσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο που επίση δεν ε, επέτυχαν. Οπότε, ε, ακόμα και, και, και αν επομένω κάποιο δεν ε, είναι υπέρ τέτοιου είδου ε, ρύθμιση επίλυση ζητημάτων, δεν υπάρχει άλλη λύση. Αυτό όμω το οποίο εμεί ε, ζητούμε, ε, και η κυρία Ρέντινγκ δεν είναι υπέρ τέτοιων λύσεων, αλλά είπαμε ότι είναι η τελευταία λύση. Θέλουμε όμω να δώσουμε την ευελιξία εφαρμογή στα κράτη-μέλη. Επίση, αναγνωρίζουμε το ότι υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα οποία έχουν ε, αναλάβει δράση στόχευμένη για το ζήτημα αυτό. Δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι παρά το ότι υπάρχουν κάποια καλά παραδείγματα, ακόμη έχουμε 15 κρατημένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα οποία δεν έχουν κάνει τίποτα σχετικά και μάλλον δεν πρόκειται να κάνουν τίποτα στο μέλλον. Επομένω, γι' αυτό θεωρούμε ότι χρειάζεται να υπάρξει μια παρέμβαση ευρωπαϊκού επίπεδου και να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ε, το ελάχιστο του σε κάθε κράτο μέλο. Νομίζω όμω ότι είναι μοναδική αυτή η οδηγία, διότι αναγνωρίζονται οι προσπάθειε που έχουν καταβάλει ήδη τα κράτη-μέλη για αυτό το ζήτημα. Επίση, τα κράτη-μέλη τα οποία δεν έχουν θεσπίσει σχετική νομοθεσία. Και έχουμε κάποια ε, καλά παραδείγματα, ε, α πούμε, στο το, το Βασίλειο, όπου με, με κουσία ρύθμιση, ε, ενδοτική νομοθεσία, ε, είχαμε αποτελέσματα. Και έχουμε και άλλα που δεν έχουν διαφερθεί καθόλου. Πάντω, εμεί αναγνωρίζουμε τι προσπάθειε που κατέβαλαν τα κρατή-μέλη, είτε προσπάθειε είναι νομοθετικού χαρακτήρα, είτε άλλου, άλλου, άλλου είδου. Ε, δεν, δεν, δεν θέλουμε να αλλάξουμε τα κράτη-μέλη δεν μας ενδιαφέρει, δεν θέλουμε να πειράξουμε κανένα κάτω μέλος. Τα αποτελέσματα ενδιαφέρουν. Αυτό θέλουμε να, πετύχουμε αυτή την πρόταση και αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντική πτυχή αυτής της οδηγίας. Οπότε και εμείς αναγνωρίζουμε τις προσπάθειες που καταβληθεί και ας τις συνεχίσουν να μελή. Επίσης φροντίσαμε να μην παρέμβουμε δυσανάλογα με τα του, του, του, του επιχειρηματικού, του εταιρικού βίου. Η πρότασή μας βασικά θέτει κάποιους ποσοτικούς στόχους. Θέτουμε αυτό το 40% για όλες τις εταιρείες. Μια εταιρεία που δεν θα πέχει το 40% δεν σημαίνει ότι θα υποστεί κυρώσεις. Εδώ έγινε μια παρεξήγηση. Τι λένε ποσοστώσεις. Ποσοστώσεις είναι για ψάρια, όχι για γυναίκες. Πολλές φορές αυτό το επιχείρημα προτάσσεται. Όχι. Αν κοιτάξετε την πρότασή μα, δεν υπάρχει λέξη ποσόστοση. Δεν θα βρείτε τη λέξη ποσόστοση. Είναι στόχο ποσοτικός το 40%. 40% των μη εκτελεστικών στελεχών στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ούτε λέμε το πώς θα το πετύχει η εταιρεία. Για μένα. Αυτό είναι το σημείο κλειδί. Το, το ανέδειξαν και κάποιοι αγορητές. Θέλουμε διαφάνεια, θέλουμε ανοιχτό πνεύμα οι εταιρείε να έχουν διαφανείς διαδικασίες επιλογής ε, με ουδέτερα κριτήρια σε σχέση με τα δύο φύλλα. Και φυσικά και υπάρχουν αρκετές ικανές γυναίκες που θα ήθελαν να έχουν μια κορυφαία θέση, στελεχική θέση. Οι οποίες οι γυναίκες τώρα από ό,τι λένε, λένε δεν έχουμε την ευκαιρία. Ποτέ δεν έχουμε διαφανή διαδικασία επιλογής. Να επομένως το βασικό στοιχείο της πρότασής μας. Τέρες που δεν έχουν το 40% τέτοιε διαδικασίες Διαφανεί θα πρέπει να υιοθετήσουν. Ούτε είναι αλήθεια ότι δεν υπάρχουν οι γυναίκες με αρκετέ δεξιότητε και ικανότητε. Εάν έχουμε υποψηφίους για μια θέση που έχουν τις ίδιες δεξιότητες, τα ίδια προσόντα, τότε είπαμε ότι θα πρέπει να ισχύσει το 40%. Και αυτό πρέπει να τονίσουμε. Μιλούμε για ισορροπία μεταξύ των δύο φύλων. Δεν μιλούμε μόνο για γυναίκες. Εάν κάποια στιγμή κυριαρχούν στη σύνθεση διοικητικού συμβουλίου οι γυναίκες, ε, τότε θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην ένταξη σε αυτό το διοικητικό συμβούλιο ανδρών. Επομένως, σημασία στη διαφάνεια. Περιορισμένη παρέμβαση στα, στα εταιρεία. Α, και κάτι άλλο πολύ σημαντικό που θα πρέπει να το τονίσω. Δεν έχω συναντήσει ούτε έναν να μου πει ότι δεν θέλουμε ισορροπία μεταξύ των δύο φίλων στην εταιρεία. Όλοι είναι πεπισμένοι ότι αυτό είναι μια ανάγκη, μια αναγκαιότητα. Ακριβώς και από πλευράς οικονομικής αποτελεσματικότητας. Όμως λένε δεν χρειάζεται να επέμβεται νομοθετικά ή να επέμβεται πανευρωπαϊκά. Όχι, να συνεχίσουν τα πράγματα όπως είναι, αυτό αποκλείεται. Προσπαθήσαμε με συστάσεις, με προτάσεις, με ενθαρρύνσεις προς τις εταιρείε για να λάβουν δράση τα κράτη-μέλη. Μερικοί το κάνανε, αλλά πάρα πολλοί δεν έκαναν τίποτα. Και για αυτό είναι σημαντικό να παρέμβουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Προτείνουμε αυτό το προσωρινό μέτρο και θεωρούμε ότι είναι σημαντικό τώρα να γίνει αυτή η αλλαγή στις νοοτροπίες, στην ουτερική κουλτούρα. Θεωρούμε όμως ότι κάποια στιγμή θα απαντήσει να χρειάζεται παρέμβαση. Και τη στιγμή ακριβώς που θα ταράξουν τα λιμνάζοντα νερά, θα έχουμε επιλογή με διαφάνεια θα έχουμε σαν, σαν ομαλή διαδικασία αυτή τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβούλιου, ε, τότε θα αποσύρουμε το νομοθέτημα. Γι' αυτό είπαμε ότι είναι προσωρινό, για να έχουμε ισότητα, δικαιοσύνη, για να υλοποιήσουμε μια από τις βασικές αξίες. Όχι, δεν είναι, δεν είναι μια σημαίνια σφαίρα. Ούτε είναι τα, τα άλλα σημαντικά μέτρα που θέλουμε να ε, έχουμε για την Είναι μια ανακοίνωση που έχουμε εκδώσει. Ε, λέμε για διάφορα μέτρα το ίδιο σημαντικά, ούτως ώστε στην πράξη να πρετανεύσει η ισότητα. Να ανάρουμε κάποια στερεότυπα, αν έχουμε ε, συμφιλίωση, να έχουμε επιλογές όσον αφορά την παιδεία, την επέκταση. Βεβαίως και τα πράγματα είναι και παραμένουν σημαντικά. Είδαμε όμως ότι όταν έχουμε ισότητα των φίλων, τότε χρειάζεται να υπάρχουν στοχευμένα μέτρα. Πέραν όλων των άλλων μέτρων που υπάρχουν για την ισότητα. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σα. Uh, well, uh, Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέροντα και πιστικά τα όσα μας είπατε. Κυρία, προφανώς θέλετε δύο λόγια για να καταλήξουμε και να δώσουμε και τα χρονοδιαγράμματα. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε ευχαριστώ τους και οδησηγητές και οδησηγήτρες που είναι παρόντες. Παρούσες εκτός από εσάς, όλες γυναίκες είμαστε. Άρα δεν έχουμε μόνο εμείς θετική στάση. Τελευταία κουβέντα λοιπόν. Η Επιτροπή με τη συμπεριφορά της μας δείχνει ότι δεν είναι απλώς πιστική η παρουσία της Επιτροπής, αλλά και η σημασία του θέματος ασφαλώς. Δεν νομίζω ότι σας επηρέασε τόσο πολύ η παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι ένα καλό παράδειγμα λοιπόν ε, αυτό. Τώρα μπορεί κάτι που ισχύει στη χώρα σας να μην ισχύει στη δική μου ή όχι σε όλες. Εν πάση περιπτώσει... Ελπίζω να μας δώσετε κι εσείς ένα καλό παράδειγμα υποστηρίζοντάς μας στην καλύτερη, μεγαλύτερη απόδοση στη δουλειά μας. Τροπολογίες στην αιτιολογήση του, της προτάσεως έχω καταθέσει. Με τη γραμματεία δεν έχω μιλήσει. Έχετε εσείς το χρονοδιάγραμμα κύριε Πρόεδρε γιατί... Ναι, λέει ο Πρόεδρος, από τα στοιχεία που έχουμε εμείς. Στέλνετε σήμερα για μετάφραση στην γνωμοδότηση, έτσι. Μάλιστα. Α, ναι, μας το αποτέλεσε. Ωραία, λοιπόν, τότε αυτό για να την συστήσουμε 11 Απριλίου στην προσοχή συνεδριαση συνεδρίαση, 5η πρωί, ελπίζω να είστε διαθέσιμοι. Το λέω. Το λέω από τώρα, συνήθω στο τέλο συνεδρίαση ανακοινώνω τη προσοχή συνεδριάσει, αλλά το λέω από τώρα, μη τυχόν και φύγει κανεί. 29 Μαου λοιπόν, εξεταστών τροπολογιών. 30 ψηφοφορία και να δούμε από εκεί και πέρα που θα πάει το θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα η συνεδρίαση. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Φαντερφλής. Χαιρετισμού θερμού στην κυρία Ρέντινγκ την οποία ιδιαίτερα συμπαθούμε στην Επιτροπή αυτή. Ήταν ενδιαφέρουσα η συνεδρίαση. Ευχαριστώ όλους όσοι έλαβαν μέρος στις συζητήσεις μας. Έχει τη σημασία του και την αξία του να κάνουμε σε κύριες, ε, σε εύστοχα και σοβαρά θέματα συνεδριάσεις. Λοιπόν, ε, μια και δεν θα ξαναειδωθούμε πριν από το Πάσχα, σε εύχομαι στους πάντες, το καθολικό Πάσχα, εύχομαι στους πάντες ε, καλές γιορτές, καλές δεκοπές, καλό Πάσχα ιδιαίτερα σε όλο το προσωπικό μας που εργάζεται τόσο σκληρά, ετοιμάζει τα έγγραφα. Ως συνήθως ευχαριστώ και τους διερμηνείς, λέει ο Πρόεδρος, ευχαριστούν και οι διερμηνείς, συμβάλλεται ιδιαίτερο και αποφασιστικά στην ποιότητα των εργασιών μας. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν 11 Απριλίου.